Okay, we are going to start the meeting tomorrow, today, this morning. Ας ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίαση. Βλέπω λιγότερους ε, παρόντες από χθες, ε, Πολύ σωστά μάντεψες. Ναι, το web streaming ίσως θέει. ναι, όχι, μάλλον ο κοροναϊός θέει. Ας προχωρήσουμε στο σημείο της ημερησίας διάταξης, έγκριση της ημερησίας διάταξης παρατηρήσεις όχι. εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη, δεν έχουμε ιδιαίτερε ανακοινώσει. πέρα από το γεγονός ότι στα εγγραφά σα έχετε την έκθεση από την ε, αντιπροσωπεία προς τη Μαδρίτη τον ε, Δεκέμβριο. Κανονική διαδικασία, αλλά πασχετός έχετε την έκθεση. Θέλετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μια παρατήρηση για τη χθεσινή συνεδρίαση. Να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής μας ε, ότι όποια και αν είναι τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φωνασκεί κανείς στο μικρόφωνο. Ε, και ε, ορισμένα μέλη απέναντι στην κυρία Τιουνμπέρκ φέρθηκαν με τρόπο καθόλου σεβαστικό και θεωρώ ότι αυτό δεν δεν είναι ε, καθόλου καλό και δεν τιμά ούτε την δημοκρατία μας ούτε περιπίτιμη ε, για το κοινοβούλιο μας. Μπορεί κανείς να μιλήσει χωρίς να φωνάζει. Ευχαριστώ. Si, si vous pensez à, à, la même personne que moi... Κοιτάξτε, ξέρω ότι υπήρχε η συνάδελφος ε, ε, η οποία πήρε την ε, θέση της συντονίστριας των ε, σοσιαλιστών γιατί ο άλλος συνάδελφος δεν δέχτηκε την θέση του και ευχαριστώ την κυρία Γιουτουρλάνδη για την θέση αυτή. Δεν υπάρχει διερμηνία, Έχετε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να τα πω αγγλικά. Just one second to say that Sylvia Έλεγα ότι η Σίλβια δεν ήταν στην ε, σωστή θέση, ε, πήρε την θέση της Γκίτουλαντ. Ε, δεν είναι σωστό, δεν είναι δικαιολογημένο, το αποφασίσαμε με την Γιούτα να το αφήσουμε γιατί δεν θέλαμε να ε, έχουμε κακή εικόνα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ την ε, Γιούτε και βεβαίως ε, θα σταλεί στον αρμόδιο κατάλληλη επιστολή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ σηκώνομαι όρθιο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω. Πρώτα απ' όλα, ο τρόπος έκφρασης ενός... Ε, ενός βουλευτή είναι ε, άσχετο από αυτό που θέλει να πει. Γι' αυτό λοιπόν η Σίλβια Σαρντόνε έχει τον ε, δικό της τρόπο. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην δικιά σας θέση. Όταν η Σίλβια Σαρντόνε τη, τελείωνε την παρέμβασή της, εσείς την υπερκαλύψατε με ένα ηχηρότατο μπλα μπλα μπλα. Η κυρία Σαρντόνε είναι και γυναίκα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ε, ε, προστατέψουμε κυρίως και τα δικαιώματα των γυναικών, άρα αυτή η στάση δεν είναι καθόλου σωστή. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος. Well, before the voting session, we need to, uh, we need to... Πριν ε, περάσουμε στην ψηφοφορία, να σας πω ποιες είναι οι συστάσεις των συντονιστών. Δεν υπάρχει καλά να περάσουμε στην ψηφοφορία. Okay, so let's start. So, amendment 38, is in favor? 38 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 δεύτερο τμήμα. Επαλήθευση. open; Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 6. 49 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση, αλλά νομίζω ότι απορρίπτεται. 49. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε μαζί ε, τις επόμενες μέχρι και την 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Uh, sorry, uh, chair, uh, Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Την ΤΕΒΕ 6 δεν πρέπει να την ψηφίσουμε.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 ε, ναι, πράγματι. Ε, πάμε πάλι. ΔΕΒΕ 6. 49. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Υπέρ. 49 μετά την ΔΕΒΕ 6. Ναι, πράγματι, ε, ψηφίσαμε την ΔΕΒΕ 6. Ε, και παραλείψαμε μία γραμμή. Πάμε πάλι. DV6, συμφωνείτε? Ωραία. DV6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Κατόπιν έχουμε την ομάδα ε, τροπολογιών υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 και 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 και 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Okay, so we go to 23 in favor. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒ1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνονται. 36 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 4 υπέρ κατά α, επαλήθευση. Δεβε 4. DV4. DV4. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. DV5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην ε, ομάδα. Προωθήσουμε το θέμα στην Ολομέλεια όσον αφορά το ε, κείμενο αυτό. Ωραία. Προχωράμε τώρα στην δεύτερη ψηφοφορία, στρατηγική προσέγγιση ε, για τα φάρμακα, ε, συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 82, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνούμε στην τροπολογία 91, υπέρ, κατά, ε, ηλεκτρονική ε, επαλήθευση επί της τροπολογίας 91 άρχεται πέρας εγκρίνεται τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 122 υπέρ κατά. Ε, καλύτερα να το ελέγξουμε. Τρόπο ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 122. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Άρα ψηφίζουμε τώρα ε, για τις 23, 24, 100, 23, 24, 25 υπέρ κατά αποχές ε, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. Τροπολογία 126. Όχι. Ναι, την ψηφίζουμε τελικά υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 126. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 132 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 132. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά να ελέγξουμε για την 146 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 147 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά προτιμώ να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την 147. Απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 171 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 171. Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Τροπολογία 172 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 173 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 180 η 181 έχει αποσυρθεί. 181 έως και 189 en bloc υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Ψηφίζουμε για την 182 υπέρ κατά αποχές Μάλλον απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Όχι πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 199 εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 203 μέχρι 205 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 208. Α, καταπίπτει 208, συμβιβαστική 15, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 212, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 καταπίπτει. Άρα φτάνουμε στη συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 237 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση απορρίπτεται 238 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 238 πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 2.39 μέχρι 2.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 242 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Επί της τροπολογίας 242 πέρας της πληροφορία απορρίπτεται. 243 υπέρ Κατά εγκρίνεται 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 245 υπέρ ποια είναι η γραμμή του ΕΛΚ κατά άρα Ναι, όταν σας βλέπω είναι και καλύτερα να, το, να δείχνετε πιο νωρίς. 245 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Και απορρίπτεται. Θα ζητούσα εκ δεξιών μου να μην, ε, να μην θορυβούν και να μην μιλούν μεταξύ τους οι αντιπρόεδροι. Πειθαρχία παρακαλώ. 246 και 247 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται όντως. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 258 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε μετά την τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 42. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία. Όχι, όχι, όχι, όχι. Πέρας της ψηφοφορίας ε, απορρίπτεται. 42 λέει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά, ε, συγγνώμη, 52 υπέρ. Όχι, να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 53 και 50 μέχρι 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Επί της τροπολογίας 63. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα ε, ψηφίζουμε την τροπολογία 65. Η 64 καταπίπτει. Άρα 65. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 65. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, αν μπορούσατε να μην βγάζετε αμέσως έτσι, τόσο γρήγορα τα αποτελέσματα από την οθόνη, να βλέπουν όλοι. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Τροπολογία 71 πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Ορίστε, τώρα το αφήσαμε στην οθόνη. Με την άνεσή σας θα διαβάσετε τα αποτελέσματα. Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 73, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 74, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 75, 75 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Νομίζω, λέει ο Πρόεδρος, ότι χρειάζομαι καφέ, δεν τα πάω καλά σήμερα πέρας της ψηφοφορίας και δίκιο είχα από την αρχή εγκρίνεται τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του κειμένου λοιπόν τώρα θα ψηφίσουμε πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται μπράβο σας και συγχαρητήρια Okay, you don't care about pesticides. Okay, so let's start again, please. Ας ξαναρχίσουμε. And we move to, uh... Περνάμε λοιπόν σε ένα ε, ζήτημα ε, αρκετά σύντομο, δηλαδή αυτό ε, που αφορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψε με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όχι το δικαστήριο, το συνέδριο, ελεγκτικό συνέδριο. Ε, το κύριο Σέμοντζερ έχει το λόγο και ξεκινάει 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή. Ε, Σα ευχαριστούμε που μα δίνετε δυνατότητα να παρουσιάσουμε την έκθεσή μα σε σχέση με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εδώ. Ε, τέσσερα κομμάτια περιλαμβάνονται. Το γιατί προβήκαμε σε αυτόν τον έλεγχο, το ποιο ήταν το φάσμα τη επιθεώρηση που κάναμε και προσέγγιση, ποιε ήταν οι παρατηρήσει μα και ποιε είναι οι συστάσει μα. Καταρχήν, ποιοι είναι οι λόγοι ε, για την διαξαγωγή αυτού του ελέγχου. Καταρχήν, έχουμε δει να υπάρχει ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον από την πλευρά του Εβραίου σε κοινό και από όμω το Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ε, και η. Ε, πωλήσει των δραστικών ουσιών ε, στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν παραμείνει σταθερέ ε, και βρίσκονται γύρω σε 400.000 τόνους ετησίω, αλλά η ε, πολλούμενη ποσότητα δεν ε, σχετίζεται ευθέω ανάλογα με ε, τους σχετικούς ε, από εκεί και μετά η οδηγία σε ό,τι αφορά την βιώσιμη χρήση ε, ισχύει εδώ και 10 χρόνια και είχε ως στόχο τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων στα, των, των φυτοπροστατικών ε, προϊόντων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Από εκεί και μετά θεσπίστηκε και η νέα προσέγγιση των ε, φυτοπροστατικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου και επίση υπάρχουν περιορισμένε ε, πληροφορίε και στατιστικέ πληροφορίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά ε, του κινδύνου. Άρα λοιπόν, ποιο ήταν το φάσμα του ελέγχου μα αυτή τη έκθεση, όχι το να δούμε ποια είναι τα φυτοφάρμακα τα φυτοπροστατικά προϊόντα που θα πρέπει να απαγορευτούν ή όχι, αλλά να δούμε κατά πόσο η ε, Επιτροπή έχει ορίσει τις συγκεκριμένε εναλλακτικέ ε, που θα χρησιμοποιούνται μετά από την απαγόρευση των ιδιαίτερα επικίνδυνων ε, φυτοπροστατικών προϊόντων και αν έχει ορίσει σχετικέ προποθέσει σε ό,τι αφορά του σχετικού κινδύνου. Άρα λοιπόν το ερώτημα ήταν αυτό. Το, δηλαδή εξετάσαμε το ποιο είναι το πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε την εξάρτηση από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και κατά ε, πόσο έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέτρα. Και ε, όλη, ο έλεγχο αυτό η έκθεση βασίστηκε στην εξέταση κειμένων αλλά και στη διεξαγωγή ε, συνεντεύξεων, αλλά και κάναμε και επισκέψει σε τρία κράτη-μέλη. Ποιε ήταν παρατηρήσει Ότι διαπιστώσαμε ότι σε γενικέ γραμμέ η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δράση για να προωθήσουν τη βιώσιμη χρήση αυτών των προϊόντων, αλλά τελικά είναι περιορισμένη η πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά τη μέτρηση αλλά και τη μείωση των σχετικών κινδύνων. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε τρει βασικού άξονε, αν θέλετε σε ό,τι αφορά αυτέ τι παρατηρήσει. Καταρχήν, η βιώσιμη χρήση των φυσιοτροφικών προϊόντων ξεκίνησε ω ε, προσπάθεια ε, πολύ αργά. Από εκεί και μετά, παρότι τι προσπάθειες έχουν γίνει, υπάρχουν λίγα κίνητρα για τους γεώργου προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή του από τα ε, φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Και τρίτον, ε, γενικότερα οι στατιστικές, τα στατιστικά στοιχεία αλλά και οι δείκτες οι οποίοι μετρούν τους σχετικούς κινδύνους και τις επιπτώσεις έχουν περιορισμένη χρησιμότητα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πρώτο κομμάτι, ε, την αργή δηλαδή έναρξη, η οδηγία για την βιώσιμη χρήση 1928 εγκρίθηκε το 2009 αλλά η ε, μεταφορά στην εθνική νομοθεσία αλλά και η εφαρμογή των σχετικών σχεδίων δράσης από τα κράτη-μέλη άργησε βέβαια, το θετικό είναι ότι από το 2016 και μετά η Επιτροπή ανέλαβε περισσότερη δράση, βλέπετε εδώ και κάποια παραδείγματα στη διαφάνεια, προκειμένου να προωθήσει την εφαρμογή αυτής της οδηγίας σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη χρήση των ε, φυτοπροστατικών προϊόντων. Ωστόσο, οι αρχικές καθυστερήσεις ε, οδήγησαν ακριβώς στο να ξεκινήσει αργά και με βραδείς ρυθμούς η εφαρμογή αυτής της ε, οδηγίας. Μετά, το δεύτερο, η δεύτερη παρατήρηση, αν θέλετε, είναι το ότι υπάρχουν λίγα κίνητρα σε ό,τι αφορά τους αγρότες και την χρήση αυτή τη ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Καταρχήν, υπάρχουν ε, εργαλεία μέσα στην κοινή γεωργική πολιτική, όπω συμβουλευτικά ε, συστήματα και ειδικά ε, προγράμματα. Άρα, λοιπόν, τα κρατη πάλι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση από την κοινή γεωργική πολιτική για να υποστηρίξουν, για παράδειγμα, ειδικότερα τη βιολογική γεωργία. Τη σήμερα ημέρα, ε, το 7% των καλλιεργούμενων ελαιών της ε, ενό αντιστοιχεί στη βιολογική γεωργία. Αλλά δεν υπάρχουν κίνητρα σε ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη φωτοπροστασία, αυτό το Integrated Pest Management, γιατί ακριβώ δεν περιλαμβάνεται κάτι τέτοιο ω προπόθεση για τη λήψη εμ, για την εκταμείευση ενισχύσεων στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική. Επίση, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ή προποθέσει που θα μπορούσαν να εμ, διασφαλίσουν ακριβώς την εφαρμογή της ε, ολοκληρωμένης πιστοπροστασίας της IPN παρότι θεωρητικά είναι υποχρεωμένοι οι γεωργοί να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές από το 2014. Η ε, Επιτροπή ανέφερε ε, το 2017 στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ότι τέτοιου είδου κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια δράση, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη. Ταυτόχρονα, ε, ε, με την ε, οδηγία για τη βιώσιμη χρήση δημιουργήθηκε και αυτή η έννοια, αυτή η κατηγορία των φυσικοπροστατικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου το 2019. Αλλά έκτοτε μόνο το 3% των όλων δραστικών ουσιών που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά θεωρούνται χαμηλού κινδύνου. Και ένα τρίτη, μια τρίτη παρατήρηση που κάναμε είπαμε ότι έχουμε λίγα στατιστικά δεδομένα. Δηλαδή διαπιστώσαμε ότι τα στατιστικά δεδομένα για τις δραστικές ουσίες ε, που δημοσιεύονται από το Eurostat δεν είναι αρκούντος ε, ε, λεπτομερή και η φυστάμενη νομοθεσία είναι πιο περιοριστική σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία και η Eurostat ε, είναι αναγκασμένη να αθρίζει τα σχετικά δεδομένα ε, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες ε, κατηγορίες. Το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να γίνει ανάλυση επιμέρους δραστικών ουσιών, για παράδειγμα, όπως τα νεοκοτινοειδή. Επίση, ε, τα δεδομένα που διαβάζονται από τα κράτη-μέλη δεν είναι αρκούντω εναρμονισμένα, γιατί τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ε, αναφέρουν τη χρήση ε, φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε καλλιέργειε και μέσα σε ε, οποιοδήποτε περίοδο, οποιοδήποτε 12 μηνών σε ευρύτερη περίοδο 5 ετών. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα μεταξύ των κρατών μελών. Η οδηγία του 2009 υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ε, υπολογίσουν εναρμονισμένου δείκτε κινδύνου και να εντοπίζουν τι τάσει που παρατηρούν σε ό,τι αφορά τη χρήση ορισμένων δραστικών ουσιών. Επίση, υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα στοιχεία προτεραιότητα. Ωστόσο, η οδηγία δεν προέβλεπε η ίδια συγκεκριμένου τέτοιου εναρμονισμένου ε, δείκτε κινδύνου. Επίση, δεν υπάρχει προστατικοποιημένο στόχο τη Ένωση σε ό,τι αφορά το κατά πόσο θα πρέπει να μειωθούν οι κίνδυνη Και επίσης ε, τα κράτη-μέλη ε, είναι ε, υποχρεωμένα να προετοιμάσουν τα εθνικά του σχέδια δράσης έχοντας ποσοτικούς στόχους, χωρίς όμως να υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Και η ποσοτικοποιημένη γενική στόχη δημοσιεύτηκαν από το, το 2018 και άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2019. Δηλαδή ουσιαστικά άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι δείκτες 10 χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. Ε, πέραν αυτού όμως οι δύο αυτοί νέοι ε, δείκτες δεν ε, λαμβάνουν υπόψη τους το πότε και το με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Με βάση λοιπόν όλες αυτές τις παρατηρήσεις κάναμε τρία, τρεις δέσμες αν θέλετε συστάσεων προς την Επιτροπή. Καταρχήν, θα πρέπει ε, τα γενικά κριτήρια τη ολοκληρωμένη φυτοπροστασία να μεταφραστούν σε πρακτικά κριτήρια που μπορούν να επαληθεύονται σε επίπεδο αγροκτήματο έτσι ώστε να συνδεθούν με τι ε, ενισχύσει τη κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 2020. Επίση, θα πρέπει ε, να βελτιωθούν τα στατιστικά που, στοιχεία που υπάρχουν για αυτά τα προϊόντα και επίση θα πρέπει να υπάρξουν καλύτεροι δείκτε κινδύνου. Και επιχαίρουμε το γεγονό το ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε πλήρω ε, ε, στο μεγαλύτερο κομμάτι τη συστάση μα, αλλά ε, δεν μα αρέσει το γεγονό ότι δεν αποδέχτηκε την σύσταση 1β, 1b σε ό,τι αφορά δηλαδή την ενσωμάτωση τη ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στην αιρεσιμότητα για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020. η IPM λοιπόν, η ολοκληρωμένη φωτοπροστασία μόνο μερικώς περιλαμβάνεται και αυτό παρότι ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν από την Επιτροπή να αλλάξει τους κανόνες της ενεργειακής πολιτικής σε ό,τι αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση ήδη για την περίοδο του 2014-2020. Πόσο μάλλον για την περίοδο μετά του 2020. Ε, αυτά από την πλευρά μου, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σαφή όλα αυτά. Θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές. Κυρία Νόβακ, Άζεκαμ. Monsieur So ah, one more, two, three, four. Okay. Good. So let's start with... Ωραία, να ξεκινήσουμε από την κυρία Μακίνες, το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέρφους ε, για την παρουσίασή τους. Αναρωτιέμαι μήπως εξετάσατε τη διαθεσιμότητα συστήματα συμβουλών προς τους γεωργούς, γιατί μια από τις μεγάλες δυσκολίες είναι η χρηματοδότηση των ερευνών, αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας ε, είναι προβληματική σε πολλά κράτη-μέλη, διότι έχουν μειωθεί οι σχετικοί πόροι. Έχετε σχετικές πληροφορίες. Ε, Συμμετείχα στις εργασίες για την οδηγία για την βιώσιμη χρήση των ε, φυτοφαρμάκων και από τις δικές μας αποφάσεις μέχρι την εφαρμογή τους ε, μεσολαβεί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακούσαμε ε, και την παρουσίαση τώρα μόλις. Νομίζω ότι μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη συμβουλών προς τους γεωργούς, διότι πολλοί γεωργοί βασίζονται στις αγροχημικές εταιρείες θα μπορούσατε να κάνετε μια ε, σύσταση ότι χρειάζονται περισσότερες συμβουλές χρηματοδοτήμονες από το κράτος προς τους γεωργούς, ώστε να ε, χρησιμοποιούν ε, συστήματα όπου να μην χρησιμοποιούν προϊόντα φυτοπροστασίας μόνο όταν είναι απαραίτητα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ε, πάλι από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον έλεγχο της χρήσης ε, των ε, προϊόντων φυτοπροστασίας και επικροτώ τους ελέγχους της χρήσης. Ε, έχετε υποβάλει πολύ καλές συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, οι Σλοβαίνοι γεωργοί και οι Σλοβαίνοι πολίτες ανησυχούν σχετικά με τους ελέγχους προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες. Λαμβάνουμε συνεχώς ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα αυτά κάτι πολύ σωστό. Αναρωτιόμαστε όμως εάν και οι άλλες χώρες ε, λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες που έχουμε για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Το θέμα αυτό συνδέεται και με τους διαθέσιμους σπόρους, όχι μόνο η έλεγχη αλλά και η η έλεγχοι είναι σημαντικοί, οι συμβουλές, αλλά και η ε, οικονομική υποστήριξη των μέτρων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. S&D, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Πώς ελέγχονται τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Ε, εμείς ε, είδαμε στην χώρα μας προϊόντα ε, μολυσμένα με ε, ουσίες απαγορευμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το όλο θέμα αυτό πώς συνδέεται με τις ενισχύσεις της γεωργίας οι σχετικές ενισχύσεις ε, στη χώρα μας είναι το μισό από ό,τι λαμβάνουν οι γεωργοί σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώ λοιπόν μπορούμε να έχουμε τα ίδια πρότυπα για τα ίδια προϊόντα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, τη βιολογική γεωργία. Ευχαριστώ κυρία Ρένα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποια ερωτήματα. Πρώτον, συμφωνώ απολύτω με αυτό που είπε η κυρία Μαγκίνες, δηλαδή ε, ότι συχνά οι ίδιε ε, οι παραγωγές εταιρείε ε, φυτοφαρμάκων συμβουλεύουν τους γεωργούς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να παράσχουν επιστημονικές συμβουλές. Επίσης, στους γεωργούς. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο αναλύει ένα χώρα με τον τρόπο αυτό μπορεί καλύτερα να καταλάβει ποιες είναι οι επιμέρους ανάγκες ε, όσον αφορά και τα βιώσιμα φάρμακα. Τρίτον, σημείο 7 της ημερησίας διατάξεως αφορά ακριβώς τις εισαγωγές. Ακούμε ότι σήμερα η Κομισιόν επιθυμεί να είναι πιο ανεκτική όσον αφορά την χρήση φυτοφαρμάκων για τα εισαγόμενα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυσκολεύονται ήδη οι γεωργοί μας να εφαρμόσουν την οδηγία. Ε, θα πρέπει η Γενική Διεύθυνση Trade να έρθει σε επαφή με την ε, Επιτροπή ε, και τις ομάδες που ασχολούνται ε, με, την, με τα φυτοφάρμακα έτσι ώστε να μην γίνουν δεκτά από την Digitrade Trade προϊόντα με που θα έχουν υποστεί τοξικά φυτοφάρμακα με φάρμακα τα οποία δεν είναι αποδεκτά. Επίσης, τι, ποια είναι η ιδέα της δέουσας επιμέλειας ε, due diligence που μπορούμε να φέρουμε εδώ για τις περιπτώσεις ε, που θα χρησιμοποιηθούν λοιπόν εναλλακτικέ δυνατότητες πριν φτάσουμε στην χρήση αυτών των ε, φυτοφαρμάκων. Άρα θα πρέπει δηλαδή να δείξουμε ποια μπορεί να είναι η δέουσα επιμέλεια των γεωργών έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά χρήση βιώσιμη. Ο κύριος ε, Χώσικ, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά αυτά που μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ε, το μεγάλο θετικό ε, είναι να μπορούμε να μπούμε σε πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις, να βλέπουμε δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις και δεδομένα για ε, τις ε, χώρες. Ε, επομένως, τα στοιχεία αλλά και η έλλειψη δεδομένων μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ακριβώς πώς έχει η κατάσταση στη χώρα τους και πώς μπορούν να βοηθηθούν κυρίως οι γεωργοί. Δεύτερον, όσον αφορά την παροχή συμβουλών στους γεωργούς, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Ωστόσο, ε, δεν χρειάζεται απλώς να βλέπουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να δούμε και να στραφούμε προς το μέλλον, τι, τι, προβλέπει η κοινή γεωργική πολιτική όσον αφορά το θέμα αυτό, γιατί εδώ χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ικανούς πόρους ε, για την αδειοδότηση ασφαλεστέρων εναλλακτικών ε, λύσεων και παροχή συμβουλών στους γεωργούς με αρκετή προβλεψιμότητα. Αυτό μπορεί να έχει πολύ καλή καλύτερο αποτέλεσμα από το να λέμε ναι, ok, συμβαίνει κάτι, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τα χρήματα, πρέπει να δούμε ε, ότι η στήριξη πλέον προς τους γεωργούς ε, πηγαίνει προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να είμαστε συνεκτικοί. Και τελευταίο όσον αφορά τις εισαγωγές, συμφωνώ και εγώ με αυτό που υπόθηκε εδώ. Έχουμε μία σαφή περίπτωση όπου δεν ε, συζητούμε μονάχα για ε, δεσμευτικές ας πούμε ε, αναφορές και κεφάλαια στις συμφωνίες. Εδώ θα πρέπει να έχουμε μία εγκάρσια αντιμετώπιση και θα πρέπει να τηρήσουμε τα ίδια ακριβώς ε, πρότυπα και στάνταρ ε, για τα προϊόντα που παράγονται εδώ και για τα εισαγόμενα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ λίγο Πρόεδρος. Από τους πράσινους έχουμε δύο ομιλητές. Thank you, Chair, and thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, λέει η κυρία Παύλους, ε, για το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, μας έδωσε πολλές ε, πληροφορίες ε, και πραγματικά τις χρειαζόμαστε αν θέλουμε να προχωρήσει η Πράσινη Συμφωνία που δεν αφορά μονάχα το κλίμα αλλά και την βιωσιμότητα και την βιοπικιλότητα. Έχω να πω κάποια πράγματα. Πρώτον, στατιστικές. Μέχρι τώρα ε, έχουμε χρησιμοποιήσει ένα σωρό ε, ανόητα που στοιχεία γιατί αν δει κανείς τα τις ενεργές ουσίες θα καταλάβει ότι η εφαρμογή των διαφόρων ε, ουσιών μπορεί να είναι ε, τελείως διαφορετικός ανάλογα με το βάρος γιατί ε, το, ο βαθμός τοξικότητας σε σχέση με το βάρος δεν είναι καθόλου όμοιος σε όλες τις ενεργές ουσίες, δραστικές ουσίες. Ε, αυτό το κάνουμε ήδη στα φάρμακα. Γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε και στα φυτοφάρμακα. Οι επίσημες στατιστικές ε, λένε ότι χρησιμοποίησαμε λιγότερα φυτοφάρμακα, αλλά στην ουσία έχουμε χρησιμοποιήσει περισσότερα ε, γιατί έχει έχουν αυξηθεί τα ε, νοικοτινοειδή, στα οποία η δραστική ουσία χρησιμοποιείται βέβαια σε πολύ χαμηλές δόσεις, γιατί ήδη σε χαμηλές δόσεις η τοξικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μετρούμε την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων στην, ε, ε, στα χωράφια μας. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε πραγματικούς δείκτες που θα δείχνουν το πραγματικό, τον πραγματικό αντίκτυπο ε, δεν θέλουμε μόνο αναλυτικές χημικές ας πούμε ε, επιβεβαιώσεις ε, σχετικά με τις δραστικές ουσίες, ε, την χρήση τους και αυτά. Θα πρέπει να έχουμε σωστή επιτήρηση της βιοπικιλότητας στις γεωργικές περιοχές. Ίσως υπάρχει κάτι, αλλά δεν συνδέεται με την χρήση των ζανιοκτώνων. γιατί εγώ έχω διαβάσει κάποια στοιχεία που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πολύ ε, έτσι ε, δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Τρίτο σημείο, προστατευόμενες ε, περιοχές. Έχουμε ας πούμε στις περιοχές Natura 2000 απαγόρευση των ε, ζυζανιοκτώνων, αλλά όχι πλήρη ε, απαγόρευση. Ε, με την έννοια ότι ο κόσμος λέει «Μα δεν υπάρχουν ζυζανιοκτώνα, δεν χρησιμοποιούνται φάρμακα σε αυτές τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000». Καθόλου έτσι δεν είναι όμως ε, και μπορεί κανείς να πάρει άδεια παρέκκλησης και εξαίρεσης που δίνεται από τις εθνικές αρχές. Επίσης, το θέμα των ε, κυρώσεων. Δεν ξέρω ε, αν μερικές φορές πρέπει να ξεκινήσει ας πούμε μία διαδικασία επιπαραβάση κατά των ε, κρατών έτσι ώστε να σέβονται τους κανόνες. Στη σελίδα 11 της δικής σας έκθεσης ε, βρίσκω μία έμεση ας πούμε έκφραση που λέει ότι η χώρα μου η Γερμανία δεν έχει ακόμα εφαρμόσει το νέο σχέδιο δράσης για τα ζενιοπτώνα. Αυτό ισχύει ή έχετε κάποια σύσταση σχετικά πώς μπορεί να αλλάξει, να διορθωθεί η κατάσταση. Και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον ε, Μάρτιν Χόιζικ που ε, ασχολήθηκε με το θέμα δεν είναι λογικό να καταργούμε, να απαγορεύουμε μάλλον τη χρήση κάποιων ζανιοκτώνων που είναι επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία στην παραγωγή της Ευρώπης και να τα αφήνουμε στην ε, εισαγόμενη παραγωγή θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε απαγόρευση ε, τροφίμων που περιέχουν ε, στοιχεία ή που έχουν υποστεί επεξεργασία ας πούμε με ε, ζυζανιοκτώνα τα οποία είναι απαγορευμένα εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Μέτσε. Ε, ευχαριστούμε πολύ και την, το Ελληνικό Συνέδριο για αυτήν την πολύτιμη νέα έκθεση. Ε, λέτε στην έκθεσή σας ότι η Κομισιόν δεν κατάφερε μέχρι τώρα να θεσμοθετήσει ε, μέτρα έτσι ώστε η κοινή γεωργική πολιτική να υποστηρίξει περισσότερο την μείωση των ζυζανιοκτώνων ποια ε, μέτρα πιστεύετε ότι θα πρέπει ε, να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει η χρήση των ζανιοκτώνων και να προχωρήσουμε σε ολοκληρωμένη ε, διαχείρισή τους και τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο φάρμα, σε επίπεδο χωραφιού έτσι ώστε να το συνδέσουμε και με την στρατηγική η οποία προβλέπεται στην, στη διαδικασία From Farm to Fork, από το χωράφι στο τραπέζι. Επίσης, δεν έχουμε αξιολογήσει σχετικά με τα ζενοκτώνα που χρησιμοποιούνται ακόμα. Μήπως όμως θα έπρεπε ε, πιο συχνά να ε, ακολουθήσουμε την προληπτική προσέγγιση, γιατί δεν το είδα στα συμπεράσματά σας. Και ε, έχω και μία τρίτη ερώτηση, η οποία αφορά την ε, αξιολόγηση των ζυζανιοκτώνων. Δεν το άκουσα στην έκθεσή σας. Ε, την αξιολόγηση, την μακροπρόθεσμη, μακροχρόνια εκτίμηση της τοξικότητας που σχετίζονται με όγκους, με την αναπαραγωγική υγεία, που σχετίζονται με την νευροτοξικότητα ή ακόμα και με τους διαταράκτες, ενδοκρινικούς διακταράκτες. Αυτή είναι η τρίτη μου ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ τον ελεγκτικό συνέδριο για αυτές τις συστάσεις που έδωσε. σίγουρα θα ασκήσουμε πιέσει από τη δική μα ε, πλευρά προκειμένου πραγματικά να αναλυφθεί η δράση σε σχέση με αυτέ τι συστάσεις. Ε, θα ήθελα όμω ε, να ε, θέσω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτού του όρου ε, της IPM, Integrated Pest Management, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Ε, στην δική μας χώρα, στις κάτω χώρες, είναι τόσο ευρία αυτή η έννοια που, για παράδειγμα, Ε, καλύπτεται και η επικάλυψη για παράδειγμα σπόρων προς ε, σπορά με νέο κοτινοειδή. Δηλαδή καλύπτει ε, πάρα πολλά διαφορετικά φάσματα χρήσης αυτών των δραστικών ουσιών. Οπότε, ουσιαστικά στη δική μας χώρα η προσπάθεια γίνεται με, με αρκετά ολοκληρωμένο τρόπο και σε ό,τι αφορά τα νέο μη ε, νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι ε, πρόκειται για βλαβερά, βλαβερές ε, χημικές ουσίες. Άρα λοιπόν ε, τέτοιου είδους ε, πρακτικές όπως δηλαδή να επικαλύπτονται με, ε, με τέτοιου είδους ουσίες ή σπόροι δεν είναι κάτι το επικίνδυνο, κάτι που δεν θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα. Ποιες είναι λοιπόν κάτι οι δικές σας γνώμη, οι δράσει οι οποίε θα πρέπει να αναλυθούν έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να έχουμε βιώσιμη ε, ε, γεωργία σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των προϊόντων. Ο κύριο Βόλα. ναι. Ε, ε, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Μαγκίνε παρότι προερχόμαστε από διαφορετικέ πολιτικέ παρατάξει. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο απολούνται αυτά τα προϊόντα είναι πολύ λανθασμένο στην Ιρλανδία. Γιατί εκείνοι οι οποίοι ε, πολλούν αυτά τα προϊόντα είναι και εκείνοι που είναι αρμόδιοι να συμβουλεύουν σε ό,τι αφορά τη χρήση του. Οπότε προφανώ θα προωθούν. Σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ε, να πω ότι ε, νομίζω πως το, ένα ελεκτικό συνέδριο αυτό μπορεί να κάνει να εξετάσει το τι έχει συμβεί στο παρελθόν και να κάνει συστάσεις από αυτού. Δεν μπορεί δηλαδή να λάβει δράση σε ό,τι αφορά το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξή. Αλλά ίσω να κάνω και κάποιο λάθο. Και από εκεί και μετά, αυτό που αναφέρει σε ό,τι αφορά την ποσοτικοποίηση, ε, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τι, το κοινό καλό, αν θέλετε. Είναι κάτι που δεν ποσοτικοποιείται. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να απομακρυνθούν οι γεωργοί μας από τα ε, φυτοπροστατικά προϊόντα, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό έχει κόστο, γιατί όταν κανεί δεν χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα, χρειάζεται να εργαστεί παραπάνω και έχει λιγότερη εσόδια. Οπότε ε, αυτό το γεγονό δηλαδή τη μειωμένη χρήση των φυτοπροστατικών προϊόντων θα δημιουργήσει περισσότερο κόστο. Οπότε θα ήθελα το ελεκτικό συνέδριο να κάνει και μια σύγκριση ανάμεσα στο αυξημένο κόστο αφενό και την αύξηση για το κοινό καλό αφετέρου. Έχουμε δηλαδή προσπάθειες που έχουν γίνει σε επίπεδο κυβερνήσεων εθνικών ε, που δεν συνοδεύονται από προσπάθειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που θέτω εγώ σε ερώτημα είναι πώς μπορεί κανείς να θέσει μια τιμή αν θέλετε για το κοινό καλό. Ε, πώς μπορεί κανείς να μετρήσει το αν και σε ποιο βαθμό κάτι είναι καλό ή όχι. Είχαμε ε, μόνο δύο μιλητέ από το ΕΛ και γι' αυτό η κυρία Μακίνης ε, θα ήθελε να ξαναπάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ξαναπάρω το λόγο. Το θέμα δεν είναι οι πολιτικές ομάδες. Προσπαθούμε να κάνουμε ε, το σωστό για τα συστήματα παραγωγή τροφίμων. Μπορεί να ε, μην ε, ανεβάζουμε πολύ του τόνου αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν πολλοί γεωργοί ε, στην Ιρλανδία και σε άλλα κράτη-μέλη, φαντάζομαι, που κάνουν γεωργία διατήρηση τη βιοπικιλότητα του εδάφου και το κάνουν αυτό επειδή του ενδιαφέρει η φύση, η παραγωγή τροφίμων και θα πρέπει να αμύψουμε αυτού που το κάνουν αυτό. Και ε, δεύτερον, ε, είχα πάει σε ε, μονάδα παραγωγής φρούτων το καλοκαίρι που χρησιμοποιούν ζωντανούς οργανισμούς για να καταπολεμήσουν τους επιβλαβείς οργανισμούς. Εμείς εκεί που δεν ε, έχουμε στηρίξει τους γεωργούς είναι στην πολιτική μας για τις εισαγωγές, ε, διότι οι γεωργοί μου λένε ωραία, απαγορεύεται προϊόντα στην Ευρώπη, αλλά γιατί εισάγεται τρόφιμα ή ε, συστατικά που χρησιμοποιούν στις ζωοτροφές που έχουν παραχθεί με τη χρήση αυτών των προϊόντων σε τρίτες χώρες. Αυτό λοιπόν δείχνει ασυνέπεια και έχουν δίκιο. Θα ήταν καλό λοιπόν ε, να, ε, εργαστούμε, να συνεργαστούμε οι πολιτικές ομάδες, να πιέσουμε τον ε, επίτροπό μας, τον Φιλ Χόγκαν. Πολλοί λένε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είναι πέρα από τον έλεγχό μας, μπορούμε μόνο να ελέγξουμε το τι γίνεται εντός της Ένωσης. Αλλά ε, εάν ε, μας ε, απασχολούν τα προϊόντα αυτά, θα πρέπει να μας απασχολεί και η χρήση τους εκτός Ένωσης. Ας ενωθούμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ η Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ. Ε, ήθελα να συμμετάσχω στη συζήτηση. Είμαι ευγνώμων που άκουσα τις απόψεις ε, συναδέλφων από διάφορες πολιτικές ομάδες που είπαν ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Θα ήθελα επίσης Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την eh, έκθεση από το Ελεκτικό Συνέδριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ε, για τον πολύ καλό διάλογο εδώ στην Επιτροπή μας. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ε, ομάδες και ότι θα μπορέσουμε έτσι να πετύχουμε αλλαγή. Δεν είναι βιώσιμη η χρήση των φυτοφαρμάκων σήμερα ούτε για τα οικοσυστήματά μας ούτε για την υγεία. Απειλείται δε και η βιοπικιλότητα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε πολύ πιο σοβαρά υπόψη μας το θέμα αυτό στο μέλλον. Χαίρομαι πολύ που ακούω ότι υπάρχει συνένεση στο θέμα αυτό. Είναι πράγματι οξύμορο το ότι επιτρέπουμε την ε, εισαγωγή προϊόντων που έχουν παραχθεί με φυτοφάρμακα που απαγορεύονται εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφενό απειλεί την ανταγωνιστικότητά μα, είναι επικίνδυνο όμω και για τα οικοσυστήματά μα. Και ε, νομίζω ότι ε, όταν ε, αναθεωρήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει και εκεί να φροντίσουμε να υπάρχουν κίνητρα για μετάβαση σε πιο βιώσιμη γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει ακόμη να ε, αντιστρέψει την κατάσταση. Ε, ε, πρέπει να το κάνουμε όμως. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή και πολύ χαίρομαι που υπάρχει συνένεση εδώ στην Επιτροπή μας. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ εγγράφομαι στον κατάλογο των ε, ομιλητών για να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το ελεκτικό συνέδριο ε, για τούτη την ε, έκθεση που και έγκαιρα έρχεται και σαφής είναι. Ε, πρόκειται για προτάσεις τις οποίες ευρέως ε, ε, συμμεριζόμαστε όχι μόνο σε τούτη την Επιτροπή αλλά και σε ένα μεγάλο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άλλωστε με την ευκαιρία της συζήτησης στην Ολομέλεια για την Πράσινη Συμφωνία Θα ξανασυζητήσαμε αυτά. Θα επανέλθω και επίσης με την ευκαιρία της συζήτησης για την πρωτοβουλία από το χωράφι στο τραπέζι From Farm to Fork ε, είναι γεγονός ότι ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς ε, τα οικολογικά σχήματα eco schemes της κοινή γεωργικής πολιτικής θα ασχοληθούν ακριβώς με αυτό το θέμα των πολιτικών δηλαδή της γεωργίας και από τη μία και τα φυτοφάρμακα από την άλλη γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε ακριβώς διασύνδεση και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και παροχή συμβουλών αλλά ε, και κινήτρων ε, και δημιουργία σωστών προϋποθέσεων έτσι ώστε να ε, κατανοήσουν οι γεωργοί περί τίνος πρόκειται. Δεύτερο σημείο, οι εισαγωγέ. Αυτό δεν αφορά βέβαια εσά τόσο πολύ όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εκπρόσωπο νομίζω της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας, DG Sante και ενδεχομένως θα θέλουν να πάρουν το λόγο με ε, καθότι γνωρίζομαι ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση ε, Γεωργίας, Εμπορίου και υγεία. Νομίζω ότι μπορούμε να ξανασυζητήσουμε με του ε, αντιστοίχου επιτρόπους έτσι ώστε να πούμε ότι υπάρχει μια τεράστια ε, ένα τεράστιο φάσμα του Κοινοβουλίου από την κυρία Μαγκίνε μέχρι τον κύριο Γουάλλα. φανταστείτε, που λένε ακριβώ το ίδιο πράγμα σχετικά με την προστασία των γεωργών και σχετικά με το τι επιτρέπεται και όχι στα εισαγόμενα προϊόντα όσον αφορά την νομική βάση. Καταλαβαίνω ότι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν ας πούμε ε, η Βραζιλία, η Ινδία ή άλλες χώρες ε, θέλουν να προστατέψουν τη βιοπικιλότητά τους, να το κάνουν. Ναι, αλλά εάν εμείς θέλουμε να πουλήσουμε αυτή την πολιτική στους γεωργούς, εάν θέλουμε να αποφύγουμε είτε την αδράνεια είτε τις συγκρούσεις, ε, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το νομικό επιχείρημα. Ε, κατανοώ βεβαίως πώς έχει το πρόβλημα ε, και κατανοώ αυτά που λέει η Γενική Διεύθυνση αλλά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε ένα προπέτασμα καπνού και να πούμε ότι α, κρυβόμαστε πίσω από εκεί και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε άλλωστε καινούργια κείμενα τα οποία θα πρέπει ε, να συγγράψουμε. Ωραία και τώρα θα ξαναβάλω το καπέλο του Προέδρου και θα τα πω στα αγγλικά και ε, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε όσον αφορά τα δικά σας θέματα και μετά θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της DG Sante. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω από την ερώτηση του κυρίου Γόλας. Τι ε, μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το κοινό καλό κλπ. Όσον αφορά τον υπολογισμό του. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θέτει το ελεγκτικό συνέδριο του στόχου, ούτε διαμορφώνει την πολιτική. Αυτά είναι θέματα ε, Κομισιόν Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το ε, ελεκτικό συνέδριο ελέγχει αν οι δράσεις που έχουν επιλεγεί ε, μας επιτρέπουν να πετύχουμε τους ε, στόχους που έχουν ε, τεθεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν δεδομένα για να διαμορφωθούν οι πολιτικές. Δεν θα μπορέσω μάλλον να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω για όλες τις απόψεις και ερωτήσεις που τέθηκαν, διότι βλέπω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ επίκαιρο το θέμα. Να ξεκινήσω λοιπόν από τις ερωτήσεις ε, της κυρίας Μακίνης σχετικά με ένα σύστημα συμβουλευτικό. Αυτό αποτελεί μία από τις ε, αρχές ε, στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και θα πρέπει να τονιστεί, αλλά εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να καθορίσουν στα εθνικά τους σχέδια τι ακριβώς είναι αυτή η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. υπάρχουν διάφορες αρχές, αλλά ε, το πώς θα εφαρμοστούν ε, θα πρέπει να είναι σαφές στις αρχές διαχείριση στα κράτη-μέλη, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουν και οι γεωργοί τι πρέπει να κάνουν για να μην ε, τιμωρηθούν. Αυτό που λέμε στην έκθεσή μα ε, είναι λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι ούτε για τον Γεωργό ούτε για τι διαχειριστικέ αρχέ, ε, διότι δεν έχουν ε, καθοριστεί σαφώ τα θέματα αυτά στα ευρωπαϊκά σχέδια δράση. Και μόλι το 2016 άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προειδοποιεί τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να βελτιώσουν τα εθνικά σχέδια δράση. όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τον έλεγχο προϊόντων από τρίτες χώρες. Έχουμε ξεχωριστό έλεγχο για τα βιολογικά τρόφιμα και διαπιστώσαμε ότι κάποιοι έλεγχοι γίνονται εξορισμού στις τρίτες χώρες, αλλά μάλλον δεν αρκούν αυτοί οι έλεγχοι και θα πρέπει να διευρυνθούν ε, ε, ώστε να μπορούν πράγματι να θεωρηθούν βιολογικά τρόφιμα από τρίτες χώρες. Λίγο πολύ την ίδια ερώτηση είχαμε και από τον κύριο Σουτάρου. Θα ήθελα να προχωρήσω λοιπόν στην ερώτηση της κυρίας Αρένα. Η ερώτησή της ήταν λίγο πολύ παρόμοια με την ερώτηση της κυρίας Μακίνες. Σίγουρα θα στηρίζαμε να υπάρχουν δημόσιοι φορείς παροχής συμβουλών, κάτι που υπάρχει εν μέρη ήδη σε κάποια κράτη-μέλη. πιο σημαντικό όσον αφορά τις εναλλακτικέ λύσεις είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι γεωργοί εάν απαγορευτούν τα φυτοφάρμακα υψηλού κινδύνου και αν υπάρχουν διαθέσιμα φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου, διότι μόνο το 3 τα 100 ε, θεωρούνται φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου μετά από πάνω από 10 χρόνια ερευνών. Ε, μάλλον λοιπόν θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά ώστε να μπορούμε να βρούμε περισσότερα ε, τέτοια φυτοφάρμακα διότι δεν αρκεί να απαγορεύσουμε κάτι, θα πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικέ λύσεις όσον αφορά την ε, ερώτηση σχετικά με τα δεδομένα σε επίπεδο κρατών μελών. Εμείς έχουμε πει ότι κάποια κράτη-μέλη όπως η Γαλλία δημοσιεύουν δεδομένα για κάθε δραστική ουσία, αλλά ακόμα και αν τα υποβάλλουν αυτά τα στοιχεία στην Eurostat, η Eurostat τα συγκεντρώνει τα δεδομένα αυτά σε υψηλότερο επίπεδο, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ε, κατάλληλες αναλύσεις. εξετάζουμε το ενδεχόμενο να παρακάμψουμε την Eurostat και να συγκεντρώσουμε τέτοια δεδομένα. Ε, σωστό λοιπόν θα ήταν να αλλάξει η νομοθεσία και να επιτρέπει στην ε, ε, Eurostat να δημοσιεύει στοιχεία για κάθε μία από τις δραστικές ουσίες ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει με την χρήση των φυτοφαρμάκων. Η κυρία Πάολους έκανε διάφορες ερωτήσεις. Η μία αφορά τις ποσότητες ε, φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται. Εμείς ε, στη δική μας έκθεση είπαμε ότι εναρμονίσαμε τους δείχτες κινδύνου και σύμφωνα με τους ε, υπολογισμούς της Κομισιόν έχει μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων κατά 20% αλλά το στοιχείο αυτό αφορά αποκλειστικά τα μη εγκεκριμένα φυτοφάρμακα και έτσι δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν αυτά οι γεωργοί. Το αν έχει μειωθεί ο κίνδυνος από τη χρήση φυτοφαρμάκων ε, δεν είναι σαφές ε, και ο δείχτης ο συγκεκριμένος ε, δεν το μετράει αυτό. Και γι' αυτό συστήσαμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τον εναρμονισμένο δείκτη κινδύνου. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω την ε, Επιτροπή ΕΝΒΗ ότι έχουμε τώρα δύο ε, ε, ελέγχους. Ο ένας έχει να κάνει με τους επικονιαστές και ο άλλος έχει να κάνει με την βιοπικιλότητα στη γεωργία στις γεωργικές εκτάσεις. Όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων σε προστατευόμενες περιοχές, αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στον έλεγχο για τους επικοινωνιαστές. Όσον αφορά τις διαδικασίες επιπαραβάση, Φυσικά θα πρέπει να βελτιωθούν τα εθνικά σχέδια δράσης ε, για να καθοριστεί συγκεκριμένα τι είναι η ολοκληρωμένη ε, διαχείριση των ε, φυτοφαρμάκων. από την άλλη, πράγματι μπορεί να επιβληθούν ποινές στους γεωργούς αν δεν εφαρμόζουν τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Στις κάτω χώρες μάλιστα είχαμε υπόθεση όπου οι αρχές διαπίστωσαν ότι το 20% των γεωργών δεν τεκμηριώνουν την χρήση φυτοφαρμάκων, κάτι το οποίο όμως είναι υποχρεωτικό. Παρ' όλα αυτά δεν επιβλήθηκαν ποινές. Τέθηκε επίσης ερώτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να ελέγξουμε τι πράγματι γίνεται στα χωράφια. Τα κράτη-μέλη πρέπει να το αποφασίσουν αυτό στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης, δηλαδή πώς μπορεί να γίνεται το έλεγχος και η επιβολή των κανόνων. Στην ε, προσέγγιση μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των εναλλακτικών λύσεων. Αυτό πρέπει να εξεταστεί πρωτού απαγορεύσουμε τα φυτοφάρμακα υψηλού κινδύνου. η κυρία Χάζεκάμπ είπε ότι στις κάτω είναι πολύ ευρύς ο ορισμός ε, της ε, ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, ε, αλλά και πάλι είναι κάτι που θα πρέπει να καθορίσουν τα κράτη-μέλη στα σχέδια δράσης τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει εάν τα σχέδια δράσης ευθυγραμμίζονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Οι υπόλοιπε ερωτήσει απευθύνονται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπω, αλλά εάν κάτι μου διέφυγε, σα παρακαλώ να με ξαναρωτήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν τα μέλη συμφωνούν, θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Σάντε, προκειμένου να κλείσει αυτή η πρώτη συζήτηση, αυτό το σημείο και μετά να ε, ξεκινήσει ε, η συζήτηση για το επόμενο σημείο τη ημέρα Σα αφού πολλά από τα ερωτήματα μέσα στα δύο σημεία σχετίζονται μεταξύ του. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην εκπρόσωπο τη Επιτροπή για να απαντήσει στο πρώτο ερώτημα και προκειμένου να μα κάνει την εισαγωγή για τη δεύτερη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη χρήση των ε, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον συνάδελφο, γιατί εκείνο είναι ο πλέον αρμόδιο και συνέχεια θα ξαναπάρω εγώ το λόγο για να κάνω την παρουσίαση για το δεύτερο σημείο. Πολύ καλά, λέει ο πρόεδρο. Καλώ λοιπόν από τα εκπρόσωπο τη Επιτροπή του. Ε, και να πούμε ε, ότι ευχαριστούμε το Ελεκτικό Συνέδριο για αυτές τις συστάσεις ε, που έκανε και ε, πράγματι έρχεται σε μια σωστή χρονική συγκυρία γιατί ένας από τους στόχους του Green Deal, της Πράσινης Συμφωνίας, είναι και ακριβώς η καλύτερη χρήση των φυτοπροστατικών προϊόντων και ποια είναι τα συμπληρωματικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και ειδικότερα από την πλευρά των χημικών φυτοπροστατικών προϊόντων. Άρα λοιπόν οι ε, ε, συγκεκριμένες δράσεις που θα προταθούν μέσα στο Green Deal σχετίζονται και με τις συστάσεις μέσα σε αυτή την έκθεση. Καταρχήν, να πούμε ότι κατά τελευταία 10 χρόνια υπήρξε σημαντική μείωση των κινδύνων που προέρχονται από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ωστόσο παραδεχόμαστε ότι περισσότερα θα πρέπει να γίνουν και περισσότερα μπορούν να επιτευχθούν. Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, το Integrated Pest Management, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που θα πρέπει να εφαρμοστεί έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτού του στόχου και προκειμένου βέβαια να εφαρμοστεί να εφαρμοστούν σε επίπεδο ε, κρατών μελών. Και εμεί ε, έχουμε συνεργαστεί στενά με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία προκειμένου να υποστηρίξουμε τη βιωσιμότητα μέσω ακριβώ τη κοινή γεωργική ε, πολιτική. Και επίση έχουμε συνεργαστεί και με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη παρακολούθηση των οικοσυστημάτων. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να καλύψω όλα τα σχόλια που έγιναν, αλλά θα αναφερθώ ε, στα βασικά μηνύματα, αν θέλετε, που προέκυψαν από τα διάφορα ερωτήματα και συνέχεια θα δώσω το λόγο στη Σαμπίνα έτσι ώστε να σχολιάσει τα ζητήματα σε ό,τι αφορά εισαγωγέ από τρίτε χώρε, ενώ θα δώσω τον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία για να απαντήσει στα όσα υπόθηκαν σε σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική. Ε, μία σειρά από σχόλια από τα κράτη-μέλη έγιναν ε, σε ό,τι αφορά την επιβολή τη νομοθεσία εδώ και την επιβολή κυρώσεων. Ε, η οδηγία ε, για την βιώσιμη χρήση ουσιαστικά αποτελεί ε, μέλος ε, της, ε, του, του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου, δηλαδή του 2017-64, που εξετάζει καταρχήν το κατά πόσο υπάρχει εφαρμογή της νομοθεσίας ή όχι. Άρα λοιπόν αυτό δίνει περισσότερες δυνατότητες στα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράσεις σε ό,τι αφορά την σωστή εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας. ε, είναι δυνατό λοιπόν μέσω ελέγχου, μέσω επιθεωρήσεων να διαπιστώνεται ο βαθμός συμμόρφωσης και η εφαρμογή της νομοθεσίας. Και θα δούμε αν πράγματι υπάρχει επαρκή συμμόρφωση και αν όχι θα δούμε κατά πόσο είναι απαραίτητη η λήψη περαιτέρω μέτρων και διαδικασιών κατά παράβαση αν χρειαστεί. Ε, μία, ένα από τις συστάσεις που έκανε ε, το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του ήταν η βελτίωση των στατιστικών στοιχείων και, των, και, και περισσότεροι δείκτες. Εμείς ήδη το είχαμε αναγνωρίσει αυτό, ότι χρειάζονται βελτίωση οι δείκτες ε, και βέβαια η ύπαρξη των δείκτων εξαρτάται και αξιοπιστέ πολύ από τα εφιστάμενα δεδομένα. Και κάναμε ε, ήδη αρκετές εκτεταμένες συζητήσεις ως προς τη συλλογή δεδομένων μέσω και ε, του κανονισμού σε ό,τι αφορά τα ε, ε, στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα φυτοποστατιστικά προϊόντα. Ε, δηλαδή, στο πλαίσιο τη αναθεώρηση τη νομοθεσία, αυτό που αξιώνουμε εμεί είναι να έχουμε μη αθροισμένα δεδομένα, ξεχωριστά έτσι ώστε να έχουμε πιο λεπτομερή δεδομένα και για τα επιμέρου κράτη-μέλη, έτσι ώστε η χάραξη τη πολιτική να γίνεται με βάση ακριβώ μεμονωμένα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και όχι αθρηστικά. Επίση, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των προϊόντων. Ε, δηλαδή, όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία μπορούμε να δούμε ε, ποιοι είναι οι δείκτες σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το βαθμό εξάρτησης, ε, το βαθμό χρήση και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βελτίωση της εφαρμογής του IPM, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, ε, η, η ανεξάρτητη δηλαδή ε, εκπαίδευση ε, και η παροχή της ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ένα ε, βήμα και ήδη υπάρχει κάτι τέτοιο ω διαδικασία, αλλά στο πλαίσιο τη αναθεώρηση τη νομοθεσία θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το βαθμό αυτονομία αλλά και το βαθμό κατάρτιση και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ό,τι αφορά το IPM, την οχρεωμένη δηλαδή φυστοπροστασία σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε δραστικέ ουσίε. Μετά, νομίζω έγινε ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά το γερμανικό εθνικό σχέδιο δράση στο πλαίσιο της προσέγγισης ε, από το αγρόκτημα στο τραπέζι έχουμε εξετάσει ακριβώς και τις δυνατότητες καλύτερης εφαρμογής της οδηγίας ε, σε ό,τι αφορά την βιώσιμη χρήση ε, των φυτοπροστατικών προϊόντων και των εθνικών σχεδίων δράσης. Το εθνικό σχέδιο δράσης της Γερμανίας έχει ήδη υποβληθεί, που αυτό σημαίνει ότι πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις αυτά και ο από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας αν θέλει να πάρει το λόγο. Από την ε, δική μας οπτική γωνία να απαντήσω Συλλογικά στις, ε, στα ερωτήματα που τέθηκαν σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, ουσιαστικά δύο είδη ερωτήσεων ε, τέθηκαν. Το πρώτο είναι με ποιο τρόπο η κοινή γεωργική πολιτική μπορεί να προωθήσει την ε, βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατικών προϊόντων από τους γεωργούς και μετά το δεύτερο ερώτημα είναι ποιε ακριβώ υπηρεσίε περιλαμβάνονται σε αυτέ τι συμβουλευτικέ υπηρεσίε για του γεωργού. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πρώτο, εμ, ερώτημα, θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην εφιστάμενη κοινή γεωργική πολιτική και τη μελλοντική. Γιατί στο μέλλον θα υπάρξουν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν προταθεί από την Επιτροπή. Πάντω, σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κοινή γεωργική πολιτική, θεωρείται ήδη ένα σημαντικό στοιχείο και η πολιτική αυτή συμβάλλει στην σωστή εφαρμογή της οδηγίας. Για παράδειγμα, μέσω της πολλαπτής συμμόρφωσης, δηλαδή σχέση ανάμεσα Στι απαιτήσει στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική και ε, την, ε, το σεβασμό τη νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Και επίση τα συμβουλευτικά συστήματα αγροκτήματο αποτελούν τμήμα τη κοινή γεωργική πολιτική, δηλαδή τα κράτη-μέλη οφείλουν να παρέχουν τέτοιου είδου υπηρεσίε συμβουλευτικέ, μεταξύ αυτών και σε ό,τι αφορά το ζήτημα ε, τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ε, και επίση σε σχέση με τι άμεσε απληρωμέ το ίδιο συμπεριλαμβάνεται και αυτή η ενημέρωση σε ό,τι αφορά την χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε σχέση και με την νομοθεσία με τα χημικά έχουμε και πάλι ε, πολύ συγκεκριμένη έμφαση σε ό,τι αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο στο πλαίσιο της κοινή γεωργική πολιτική. Υπό τον πυλώνα 2 έχουμε συγκεκριμένε χρηματοδοτικέ ε, δυνατότητε σε ό,τι αφορά δηλαδή κλιματικέ και υπεραλωτικέ δράσει και εδώ περιλαμβάνονται ε, ε, τα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε δράσει που μπορούν να χρηματοδοτηθούν όπω η έρευνα, ε, συμβουλέ κατάρτιση και ούτω Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μελλοντική την υγειολογική πολιτική, θέλουμε να ενισχύσουμε περισσότερο την συμβολή της στην τήρηση της νομοθεσίας. Δηλαδή, η μελλοντική οι μελλοντικές ερωσιμότητες θα περιλαμβάνουν την, όλες τις διατάξεις αυτής της οδηγίας και θα επιτρέπουν την ε, συσχέτιση ακριβώς αυτής της, α, της αιρεσιμότητας συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά δηλαδή την οδηγία για τα αυτοπροστατευτικά με την εκταμείευση των άμεσων πληρωμών. Και αυτό βέβαια ε, θα ασκήσει τις πιέσεις στους γεωργούς για να εφαρμόσουν σωστά αυτές τις διατάξεις γιατί θα υπάρχει ακριβώς αυτό ο κίνδυνος του να μειωθούν οι άπρεστες πληρωμές τους. Από εκεί και μετά θα υπάρξουν συμπληρωματικά μέτρα, κίνητρα. Ε, για παράδειγμα αναφερθήκατε ε, στο, ε, στα eco schemes και πράγματι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το κονδύλι από τον πυλώνα 1 σε ό,τι αφορά ακριβώς την καλύτερη χρήση των φυτοφαρμάκων για την προστασία των ε, ε, οικοσυστημάτων. Από εκεί και μετά υπό τον πυλώνα 2 είπαμε ότι θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες ευελιξίας για τα κράτη-μέλη και στα ε, σχέδια δράσης τους τα κράτη-μέλη δράση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα προβλέπουν στρατηγική συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τη, χρήση, τη βιώσιμη χρήση των φαρμάκων. Άρα λοιπόν θεωρούμε πως με αυτόν τον τρόπο υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουμε περαιτέρω την ε, βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν των ε, νομιμοθετικών μόνο υποχρεώσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τις βουλευτικές υπηρεσίες και τα ερωτήματα που τέθηκαν, πράγματι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι γεωργοί δηλαδή χρήζουν ε, συμβουλών έτσι ώστε να εφαρμόσουν τις σωστές πρακτικές σε ό,τι αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων η υπηρεσία, η τρέχουσα υπηρεσία, συμβουλευτική υπηρεσία προς τους γεωργούς, ήδη περιλαμβάνει ένα τέτοιο στοιχείο. Δηλαδή, οι γεωργοί τη σήμερα ημέρα στο πλαίσιο τη τρέχουσα κοινή γεωργική πολιτική έχουν το δικαίωμα να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν συμβουλέ από την Εθνική Αρχή σε ό,τι αφορά και την βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Και πώ βέβαια κάτι τέτοιο αξιολογείται και εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη, ρώτησε η κυρία εμείς ε, ε, εκπονούμε αυτή την περίοδο μία μελέτη σε σχέση με ακριβώς αυτό το ζήτημα και θα έχουμε τα αποτελέσματά της ε, σε ένα μήνα. Και βρισκόμαστε σε συζήτηση με τα κρατημήλια, έχει ήδη προβλεφθεί ένα workshop για φέτος και ήδη υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μια συμβουλευτική υπηρεσία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Ναι, η κυρία Αρένα τώρα για το ερώτημα που έθεσε να πω, κλείνοντα σε ό,τι αφορά δηλαδή τον ουδέτερο χαρακτήρα, τον αμερόληπτο χαρακτήρα ε, των συμβουλών που δίνονται. Αυτό ήδη το εγγυάται το, το σύστημα όπως έχει δημιουργηθεί, το σύστημα δηλαδή παροχή συμβουλών προ του γεωργού. αλλά από εκεί και μετά θα βασιστούμε και στην δική σα υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να διασφαλίσουμε την αμεροληψία αυτών των συμβουλών. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και θα ασχοληθώ με τις ερωτήσεις, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, να σας δώσω μια γενική έποψη του που βρισκόμαστε όσον αφορά την αξιολόγηση των κανονισμών για τα ε, ζανιοκτώνα. Έχουμε ανοίξει διάφορα πεδία εργασίας, έχουμε την Πράσινη Συμφωνία μαζί με την στρατηγική από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες, τις επόμενες εβδομάδες. Ε, επίσης ε, θα έχουμε την ε, αξιολόγηση του REFIT και τη δεύτερη έκθεση όσον αφορά την αξιολόγηση για την οδηγία για τη βιώσιμη χρήση. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνδέσουμε τους ε, στόχους ε, με τα διάφορα στοιχεία της Πράσινης Συμφωνίας. Η έκθεση REFIT προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί πλήρως με την αξιολόγηση, ε, μελέτη αξιολόγησης της REFIT και θα λάβει υπόψη τον προβληματισμό που εξέφρασε μέσω δύο ψηφισμάτων ε, το Κοινοβούλιο σχετικά με τις ε, αδειοδοτήσεις και σχετικά με τα ζυζανιοκτώνα. λαμβάνουμε υπόψη είναι ότι το Κοινοβούλιο γνωρίζει ότι έχουμε διαδικασία αδειοδότησης πολύ αυστηρή. Ωστόσο υπάρχει κάτι που πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό είναι η ε, υλοποίηση και η αποτελεσματικότητα σχετικά ε, με τον τρόπο με τον οποίο ε, υλοποιούμε, εφαρμόζουμε τον κανονισμό. Αφενός λοιπόν επιβεβαιώνουμε ότι ε, οι κανονισμοί αποτελεσματικά προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή ε, και όλα τα κριτήρια έγκρισης είναι πολύ αυστηρά και παρακαλώ να σημειώσετε ότι το ποσοστό ενεργών ε, ουσιών ήδη είναι, δραστικών ουσιών είναι ήδη πάρα πολύ ε, χαμηλό για πολλές δραστικές ουσίες ε, και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό αποτελεί αντικείμενο ε, της ε, περαιτέρω εργασίας που πρέπει να γίνει μαζί με την προσπάθεια ε, μείωσης της εξάρτησης από χημικά ζυζανιοκτώνα. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι δράσεις που θα πρέπει να ληφθούν και τα μέτρα θα αφορούν αυτήν την βελτίωση καθώς επίσης και τη βελτίωση της διαφάνειας. Άλλωστε υπάρχει και το κείμενο σχετικά με την διαφάνεια και βιωσιμότητα του συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προβλέπεται σειρά δράσεων που θα, αντιδράσει, που θα αντιμετωπίσει ακριβώς τα κύρια ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την διαδικασία αξιολόγησης REFIT ε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, όπως είπα και την μείωση της εξάρτησης από τα χημικά ζυζανιοκτώνα. Όσον αφορά τις ερωτήσεις, ακούσαμε από το συνέδριο ότι αυτή τη στιγμή οι ε, δραστικές ε, ουσίες ε, χαμηλής περιεκτικότητας αποτελούν το 3% του καταλόγου των δραστικών ουσιών. Η Κομισιόν έχει ήδη αναλάβει δράση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα αλλά και τον καθορισμό τέτοιων ουσιών χαμηλού κινδύνου. Αυτό βέβαια συνδέεται και με τις καθυστερήσεις στο σύστημα αναθεώρησης ε, που αυτή τη στιγμή εντοπίζονται στα κράτη-μέλη γιατί ξέρουμε ότι ε, πολλές από ότι λίγες είναι οι ε, ε, ουσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν αλλά που θα, και θα ελεγχθούν θετικά αλλά θα πρέπει να περάσουν από αυτήν την διαδικασία ελέγχου. Επίσης έχουμε περίπου 10 νέες αιτήσει κάθε χρόνο. 50% από αυτές αφορούν ουσίες οι οποίες αναμένονται ε, να είναι χαμηλού κινδύνου ή βιολογικές αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία ε, και οι σχεδιαστές των, των ε, ε, γνωρίζουν ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση για το μέλλον. Ναι, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία, ωστόσο ευτυχώς το μέλλον δεν είναι τόσο κακό. Το μεγάλο ζήτημα βέβαια σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα Ίσως θα πρέπει να σας εξηγήσω το εξής. Το βασικό επίπεδο καταλήπων, το MRL, είναι ένα επίπεδο το οποίο ε, δεν αλλάζει. Είτε μιλάμε για προϊόντα τα οποία παράγονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ή εκτός και εισάγονται επομένως. Πρόκειται για ένα επίπεδο το οποίο έχει αξιολογηθεί από άποψη κινδύνου, έχει καθοριστεί βάσει συγκεκριμένων ε, ε, μελετών που έχουν γίνει από την ΕΦΣΑ και είτε πρόκειται για εισαγόμενα, είτε πρόκειται για ε, εσωτερικώς παραγόμενα προϊόντα, η αξιολόγηση είναι η ίδια. Και επομένω, από άποψη προστασία τη υγεία των καταναλωτών, δεν υπάρχει καμία έλλειψη συνοχή όσον αφορά την αντιμετώπιση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δραστικές ουσίες είτε δεν έχουν εγκριθεί ε, αρχικά στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να συμβεί ας πούμε γιατί δεν υπάρχει σχετικό αίτημα ή ε, μπορεί γιατί η Ευρώπη έχει άλλους επιβλαβείς επιβλεβεις από ότι άλλα μέρη ε, του κόσμου άρα δεν χρειάζεται να υπάρξει αίτημα διοδότησης είτε γιατί δεν έχουμε τέτοιες σοδιές για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί αυτό το φυτοφάρμακο. Ε, υπάρχουν όμως και δραστικές ουσίες τις οποίες απαγορεύουμε και όταν τις απαγορεύουμε το MRL είναι χαμηλότερο ε, και εν πάση περιπτώσει είναι το χαμηλότερο αποδεκτό MRL το οποίο θα εφαρμοστεί ε, και στα εισαγόμενα προϊόντα. Έχουμε ακούσει πολλά για, ε, και γίνεται πολλή λόγος για ίσες δυνατότητε ανταγωνισμού. Όταν μιλάμε για εισαγωγές ε, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς εισάγουμε. Εισάγουμε πολλά τα οποία και εμείς παράγουμε στην Ευρώπη, αλλά εισάγουμε και προϊόντα και αγαθά τα οποία δεν παράγονται ε, στην Ευρώπη ή τα παράγουμε σε ανεπαρκή ποσότητα κάποια εξωτικά φρούτα, κάποια ε, ας πούμε καφές, ε, τσάι και ε, κάποια ειδικά λαχανικά μπορεί να είναι τέτοιου είδους προϊόντα. Επίσης ζωοτροφές αυτή τη στιγμή ιδιαιτέρως εξαρτώμεθα και σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλιστα από εισαγωγές κυρίως όταν μιλάμε για τη σόγια. Επομένως ένα πράγμα είναι η η ε, ε, ίση όρια ανταγωνισμού, από την άλλη πλευρά όμως και μια άλλη συζήτηση είναι το θέμα της εξάρτησης. Και εξήγησα ε, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών τα οποία εισάγουμε. Βεβαίως η ανθρώπινη υγεία είναι το κύριο μέλημά μας και δεν είναι πιο ανεκτική η Κομισιόν για τα πολύ τοξικά ε, ζυζανιοκτώνα. Δεν είναι σωστό να λέει κανείς κάτι τέτοιο. Εάν ε, τα ζυζανιοκτώνα είναι πολύ τοξικά, ε, δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να υπάρξει MRL ασφαλές. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε τιμή μέγιστου επιτρεπόμενου καταλήπου. Ε, τώρα, η έλεγχη. Ήδη εξήγησε ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου ότι ε, στην οργανική παραγωγή γίνεται έλεγχος, επίσης ε, γίνονται έλεγχοι και στις τρίτες χώρες μετά από αιτήματα ε, σχετικά με την εφαρμογή συγγνώμη, των ζανιοκτώνων, τα σχετικά συνοδευτικά, σχετικές συνοδευτικές εκθέσεις είναι δημόσια διαθέσιμες και επομένως μπορεί κανείς να δει με ποιο τρόπο γίνονται οι έλεγχοι και με ποιο τρόπο οι αιτήσει για τα να μελετώνται. Επίσης γίνονται έλεγχοι ε, σε επίπεδο εισαγωγών. Υπάρχει μία σειρά αγαθών που υφίστανται ενισχυμένο συνοριακό έλεγχο και όπου ελέγχεται αναλυτικά και μετράται ε, ο βαθμός καταλήπων ε, φαρμάκων ζενιοκτώνων. Τέλος, έχουμε και εκτεταμένους ελέγχους της αγοράς ε, αναλύουμε 80.000 δείγματα που αφορούν και εισαγόμενα και εσωτερικώς παραγόμενα προϊόντα. Πρόεδρος, ε, δυστυχώς θα πρέπει να σας σταματήσω εδώ γιατί έχουμε ακόμα 10 λεπτά στην διάθεσή μας ε, και θα ήθελα να δώσω και κάποιο χρόνο στην, ε, στα μέλη της Επιτροπής, όχι μόνο στην Κομισιόν. Λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας όσον αφορά τους αγορητές από πλευράς Κοινοβουλίου. That's it. Okay. I close the list. Okay. Yeah, okay. So we... Ωραία, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με εσά γιατί εσείς συζητήσατε τον λόγο. Η κυρία Πάολου, ε, σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο 10 λεπτά μας έχουμε μείνει. Δύσκολο λοιπόν το έργο μου αλλά θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό για μένα θέμα. Ε, υπήρχε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πέρσι και ο λόγος ήταν ότι ε, διάφοροι παραπονέθηκαν ότι η Οδηγία 11.07 δεν προστατεύει επαρκώς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, διότι μόνο διότι οι δραστικές ουσίες ε, ε, ελέγχονται μόνο στο πλαίσιο των ε, σχετικών οδηγιών και κατευθυντηριών γραμμών, αλλά δεν επιλέγει μια επιχείρηση ποια είναι η δραστική ουσία και ποια όχι. Τα κράτη-μέλη που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των προϊόντων μπορεί να πούν ότι άμα δεν ελέγξατε τη συγκεκριμένη ουσία, η οποία είναι πολύ σημαντική. Έτσι, τα κράτη-μέλη μπορούν εύκολα να πούν ότι Είπατε ότι ε, το θεοκλαπρίτη είναι η δραστική ουσία, μπορεί να υπάρχουν ε, και άλλες. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, δώστε μας τα απαραίτητα στοιχεία. Από ό,τι γνωρίζω όμως τα κράτη-μέλη ποτέ δεν κάνουν κάτι τέτοιο, τα μείγματα δεν εξετάζονται σωστά και θα ήθελα να ρωτήσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο σκοπεύει να το διασφαλίσει αυτό και να θεσπίσει οι κανόνες για το σωστό έλεγχο των προϊόντων και όχι μόνο των δραστικών ουσιών, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, όλες οι ουσίες που περιλαμβάνει ένα προϊόν φυτοπροστασίας ε, ε, μπορούν να ε, ενισχύσουν την τοξική ενέργεια του προϊόντος. Επίσης, σκοπεύεται στην 11.07 να εισάγεται κάποια από τα στοιχεία της σχετικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι έδειξε η αξιολόγηση ε, αυτής της έκθεσης, ε, διότι αλλιώς ε, με τα νεονικοτινοειδή μπορεί να δούμε καταστροφικές συνέπειε. Δέκα λεπτά μας μένουν μόνο, οπότε θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ΕΛΚ, η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες ερωτήσεις. Η μία σχετίζεται με τα επίπεδα επενδύσεων ε, στην έρευνα και καινοτομία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ε, επιχειρήσεις που ε, παράγουν τέτοια προϊόντα δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων προϊόντων λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος ελέγχου που απαιτείται μέχρι να διατεθεί στην αγορά το προϊόν. Και δεύτερον, ε, όλοι γνωρίζουμε ε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει καταστροφή από ακρίδες σε πολλές ε, αφρικανικές χώρες. Χρειάζεται να έχουμε ισορροπημένη ε, εικόνα σχετικά με τη χρήση αυτών των προϊόντων αυτών, ε, διότι υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις ε, και θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτηση από, τις, από τα προϊόντα αυτά. Πολύ θα με ενδιαφέρε να μάθω πώς μπορούμε ε, να βελτιώσουμε τη διαδικασία, όχι μόνο να γίνει πιο γρήγορη, αλλά να έχουμε και πιο καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε ότι η μείωση της χρήσης των ε, φυτοπροστατικών ε, προϊόντων αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια. Αυτό ισχύει και γνωρίζουμε ταυτόχρονα όμως ότι τα επίπεδα καταλήπων σε διάφορα τρόφιμα στην Ευρώπη βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από πουδήποτε στον κόσμο. Και από εκεί και μετά να πω σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, ότι ε, ε όντας ουδέτερο, ότι ε, δηλαδή πραγματικά περισσότερες ε, επιχειρήσεις από το τομέα της γεωργίας κινούνται όλο ένα και περισσότερο προς την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι δεν μπορεί να υφίσταται χρήση τέτοιου είδου προϊόντων. Οπότε το δικό μου το ερώτημα είναι το εξή. Υπάρχουν εμ, διαφορετικές ε, περιπτώσεις έκτακτων, αν θέλετε, εγκρίσεων και υπάρχουν, για παράδειγμα, και συγκεκριμένα, εμ, συγκεκριμένες ουσίες οι οποίες ε, χρησιμοποιούνται σε ορισμενα κρατημένα, οπότε θα θέλαμε να ξέρουμε πώς αυτά λαμβάνονται υπόψη της εργασίες των κρατών μελών. Ευχαριστώ, ε, κύριο Σαπόλσακ. Ε, θα είμαι σύντομος. Πρέπει να αναλογιστούμε το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις μέσω, για παράδειγμα, της έρευνας, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν ε, διάφορα, διαφορετικά εναλλακτικά προϊόντα. Γιατί βέβαια ε, η ανάπτυξη τέτοιων διαφορετικών ε, προϊόντων ε, απαιτεί μεγάλο κόστο ε, και είναι μια δύσκολη διαδικασία. Άρα το ερώτημα μου προ την Επιτροπή είναι πώ μπορούμε να δώσουμε μια, ένα κίνητρο για την ανάπτυξη τέτοιων εναλλακτικών προϊόντων. Γιατί νομίζω πω υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε ό,τι αφορά εναλλακτικά, πιο φιλικά προ το περιβάλλον δηλαδή, φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Και από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των υφιστάμενων δεδομένων, ε, σε ό,τι αφορά την τοξικότητα και την αποτελεσματικότητα των ε, ε, προϊόντων αυτών, θα πρέπει η να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για όλα τα κράτη-μέλη αλλά και τις επιχειρήσεις. Η κυρία Ρένα, ευχαριστώ πολύ. Είπαμε και προηγουμένως ότι όσον αφορά το θέμα των ε, ορίων των τοξικών ε, καταλήπων. Ε, είπατε ότι είναι ακριβώς ίδιο και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο για τα εσωτερικώς παραγόμενα και τα εισαγόμενα. Ωστόσο, έχουμε εδώ μια έκθεση σχετικά με κάποια στοιχεία όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί για αυτό που κάνετε όσον αφορά την τροποποίηση για τα τοξικά κατάλοιπα ε, σε τρόφιμα. Απ' την άλλη μεριά ε, υπάρχουν παραγωγές όπως η μπανάνα ας πούμε ε, που χρησιμοποιούν πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό χρήσης ζυζανιοκτώνων που ναι δεν έχουν κατάλοιπα αλλά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην βιοπικιλότητα. Άρα το πρόβλημα είναι στη βιοπικιλότητα σε αυτή την περίπτωση. Τρίτον, ξέρετε, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους ελέγχους και στις δημόσιες υπηρεσίες και στους ελέγχους στα σύνορα. Ξέρουμε όμως ότι ε, είναι ελλειπής η πόρη όσον αφορά ε, το, τις εισαγωγές. Ας πούμε, στην Αμβέρσα ε, είναι το λιμάνι ε, από το οποίο περνούν ε, κορμί δέντρων με παράνομο τρόπο. Εγώ ασχολήθηκα λοιπόν με, αυτή, με αυτό το θέμα της ξυλίας. Εάν περνούν ολόκληρη κορμί δέντρων. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τον ελληπή έλεγχο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταλαβαίνω τι εννοείται όταν λέτε έλεγχο στα σύνορα, αλλά πρέπει να επαγρυπνούμε όσον αφορά ε, την τοξικότητα γιατί υπάρχουν ελλείψεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σπυράκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος στόχος ε, της ε, γεωργίας ε, δυστυχώ είναι η μεγιστοποίηση τη παραγωγή προκειμένου να μεγιστοποιήσουν οι παραγωγοί τα κέρδη του. και ένας από του τρόπου τη μεγιστοποίηση τη παραγωγή είναι ακριβώ η χρήση των φυτοφαρμάκων με αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβάλλοντο αλλά και τη ανθρώπινη υγεία, όπω έχει αποδειχθεί από επιστήμονε αλλά και με κυβερνητικέ οργανώσει. Ε, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δηλαδή ε, εισφραίουν μέσα στα υπόγεια έδατα και έχουν αρνητικό αντίκτυπο ε, στην πανίδα, δηλαδή σε ηχθείς, σε έντομα, σε πουλιά και αυξάνουν το κίνδυνο για τους καταναλωτές αλλά και για τους ίδιους τους γεωργούς. Άρα λοιπόν, ένα, από τα, ένα ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι το εξή. στην προσέγγιση από το αγρόκτημα στο τραπέζι, ένα από του στόχου είναι να έχουμε υγιή τρόφιμα, ναι, ασφαλή δηλαδή ε, τρόφιμα. Οπότε ε, σε αυτό το πλαίσιο θέλετε να ε, έχετε ένα αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιπτώσεων αυτών των προϊόντων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ε, ίσως να θυμόσαστε ότι υπήρξε και ένα εργαστήριο για παράδειγμα το οποίο ε, χρειάστηκε να κλείσει επειδή ε, κατηγορήθηκε ότι ε, έκανε δοκιμές σε ζώα και θεωρήθηκε δηλαδή ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών του δεν ήταν αξιόπιστα. Ευχαριστώ. Ε, θα ξεκινήσω από κάτι απογοητευτικό. Το, ε, η έκθεση για το REFIT που υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από ένα χρόνο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη. Τώρα έχουμε αυτό το πολύ ε, βαρύ έγγραφο το οποίο είναι η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. που δίνει σαφή εικόνα, λέει ότι δεν είναι πολύ καλός ο τρόπος ε, που εφαρμόζεται η οδηγία αυτή τη στιγμή και δεν ε, μας προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Υπάρχουν πρωτοβουλίες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είδαμε ότι θα υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες για να επιταχυνθεί η αδειοδότηση εναλλακτικών προϊόντων καθώς και της βαθμιαίας απόσυρσης προϊόντων αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω τα εξή. Ε, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι το 50% των αιτήσεων ε, αφορούν ε, φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου. Για μένα είναι σαν να ακούω ότι από τις νέες πηγές ενέργειας το 50% είναι ανανεώσιμες. Όχι, 100% χρειαζόμαστε στη διαδικασία αδειοδότησης και πώς θα το πετύχουμε αυτό. Πώς θα επιταχύνουμε τη διαδικασία. Και τι θα κάνουμε με την ε, αδειοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 17. Ε, βλέπουμε παράταση της ε, διάρκειας ε, της άδειας φυτοφαρμάκων που έχουν ιδιότητες που δεν θα επιτρέψουν την αδειοδότησή τους στο μέλλον. Παρόλα αυτά παρατείνεται η αδειοδότησή τους. Νομίζω ότι επιγόντως θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Πράσινη. Οι κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν δείχνουν ότι δεν προστατεύουν επαρκώς το περιβάλλον και ένας λόγος είναι ότι αναπτύσσονται σε συνεργασία με την βιομηχανία και όχι με πανεπιστημιακούς και Γι' αυτό απαιτείται αξιολόγηση κινδύνου των προϊόντων αυτών για να αποφύγουμε την απώλεια βιοπικιλότητας. Ε, Μάλιστα γνωρίζουμε ότι υπήρξαν απάτες όσον αφορά τα, τις δοκιμές ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, αναθεωρεί τα ισχύοντα ε, έγγραφα μαζί με επιστήμονες και όχι με τις επιχειρήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί επίσης ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίσει ανεξάρτητη αξιολόγηση ομοτήμων και ότι αυτή αποτελεί αξιόπιστη πηγή ε, γνώσεων στη διαδικασία αυτή. Αναγνωρίζει ότι οι ε, δοκιμές που ε, χρηματοδοτούνται από, την, από το σχετικό βιομηχανικό τομέα από εξορισμού είναι προβληματικές. Επίσης ε, τέθηκε ήδη ερώτηση σχετικά με τα καρκινογενή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Χάζεκάμπ, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήταν ε, ωραίο αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση που έθεσα πριν στο ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με τις επιστρώσει των σπόρων. Επίσης, τι μέτρα θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διασφαλίσει οι δοκιμές αυτές να αφορούν και ε, τοξικότητα σε βάθος χρόνου, όπως είναι οι καρκινογενείς, ε, τα καρκινογενή αποτελέσματα ή οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Ε, επίσης, όσον αφορά την παράταση κατά ρουτίνα των κάποιων προϊόντων, τι γίνεται, διότι εμείς είχαμε θέσει το θέμα αυτό πριν αρκετά χρόνια, ε, φαίνεται να μην έχουν συμβεί πολλά στον τομέα αυτών, ε, διότι παρατείνει την άδεια για 34 ουσίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αναφερθεί ο φόρτος εργασίας ε, του ΕΦΣΑ γιατί δεν ε, εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το άρθρο 21 ακόμα και για ουσίες ε, που ε, εξετάζει η ΕΧΑ. Επίσης το 2010 είχαμε ουσία που εκ των υστέρων θεωρήθηκε τοξική. Αυτό το τοξικοναζόλ μπορείτε να μας πείτε τι καθεστώς έχει μετά τη συζήτηση στη ΣΚΟΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι παραπάνω διότι έχουμε να συζητήσουμε τον κοροναϊό και έχετε πολλές ερωτήσεις να απαντήσετε που αφορούν και τη στρατηγική ε, από το χώμα στο τραπέζι του καταναλωτή ουσίες οι οποίες δεν είναι δραστικές. Κατανοώ αυτά που λέτε ε, για τα μείγματα. Ε, ναι, προχωράει ε, η εργασία αυτή. Και στην Μόνιμη Επιτροπή ΝΑΤΣΕ συζητούμε το θέμα αυτό και λαμβάνουμε υπόψη τις συνέργειες. Όσον αφορά δε τα μείγματα και η ΕΦΣΑ έχει προχωρήσει πολύ. Περιμένουμε δύο τελικές εκθέσεις τον μήνα Απρίλιο για τα μείγματα. Το ένα ε, αποδεικνύεται ιδιαίτερα περίπλοκο από επιστημονικής ε, πλευράς. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο από επιστημονικής απόψεως να αποφασίσει κανείς βάσει των δύο συστημάτων. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τον Απρίλιο θα μας τα πει η ΕΦΣΑ. Η μείωση της εξάρτησης συμφωνώ απολύτως. Αυτό είναι ο στόχος μας παντού. Πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση, πρέπει να έχουμε γεωργούς που θα χρησιμοποιούν ε, το σύστημα ολοκληρωμένη διαχείρισης ε, ζυζανιοκτώνων. Έχουμε εργαλεία έτσι ώστε να εξηγήσουμε πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Ε, όσον αφορά τους επικαλυμμένους πόρους, ναι, ε, είναι ένα ε, συγκεκριμένο ε, γεγονός, δηλαδή αν επικαλύψεις τους σπόρους ως μέθοδος, ναι, μπορεί να παρουσιάσει πολλά πλεονεκτήματα και σε σχέση με τη χρήση νέων οικοτινοειδών. αλλά ε, παρ' όλα αυτά ε, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή. Ε, βιολογική καλλιέργεια χωρίς ζυζανιοκτώνα. Ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε πολλές, πολλές, πολλούς περιορισμούς όσον αφορά το θεϊκό χαλκό και θέλουμε ε, και σε αυτή την περίπτωση να βοηθήσουμε την, στην μείωση ε, της χρήσης ε, φαρμάκων στη βιολογική καλλιέργεια, γιατί και αυτοί έχουν δικά τους προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αντι, ανάπτυξη χαμηλής επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων, ζανιοκτώνων, ναι, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει αρχίσαμε να αναθεωρούμε τις απαιτήσεις στοιχείων και δεδομένων έτσι ώστε ε, τα αιτήματα της ε, ε, βιομηχανίας να είναι πολύ συγκεκριμένα και απολύτως σε σχέση με το υποανάπτυξη προϊόν. Θα τα δούμε βέβαια και αργότερα ξανά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, εγώ μπορώ να περιμένω. Την άλλη μεριά καταλαβαίνετε ότι έχουμε ε, άντε πόρτα ε, την Πράσινη Συμφωνία, άρα κάπως θα πρέπει να ενταχθούν όλα αυτά σε αυτήν. Ευχαριστούμε την Επιτροπή την... και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή, ο Επίτροπο και η Γενική Διεύθυνση Υγείας θα μελετήσει ενδελεχώ το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ όλου και θα περάσουμε τώρα στο επόμενο και τελευταίο σημείο της ε, σημερινή μας ε, συνεδριάσεως ε, αφορά τον κορονοϊό. Έχω δύο ομιλητέ εδώ, πάλι εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΤΕ, ο κ. Ράιαν, και έχουμε και έναν ομιλητή από την Στοκχόλμη σε τηλεδιάσκεψη. Ελπίζω ότι τα τεχνικά συστήματα θα λειτουργήσουν. Είναι διευθύντρια της ECDC Η κυρία Άμον θα είναι λοιπόν σε τηλεδιάσκεψη από την ε, Στοκχόλμη. Ο κύριος Ράιαν 10 λεπτά για να μας πει πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές από την Κομισιόν. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχέση με την κατάσταση που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Οι Υπουργοί Υγείας συνήλθαν για πρώτη φορά στις 13 Φεβρουαρίου για να συζητήσουν ε, αυτή την ε, περίπτωση προκειμένου να συντονιστεί και η ετοιμότητα. Ε, και τότε υπήρχαν δηλαδή το Φεβρουάριο 34 περιπτώσεις που είχαν αντοπιστεί στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τρεις εβδομάδες λοιπόν αργότερα έχουμε 3.400 κρούσματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μονακό, το Σαν Μαρίνο και η Ελβετία περιλαμβάνονται μέσα σε αυτές τις χώρες. Βλέπετε λοιπόν ε, την διαφορά ανάμεσα στα 44 κρούσματα αφενός και 3.400 κρούσματα αφετέρου. Τα περισσότερα βέβαια από αυτά βρίσκονται στην Ιταλία, 2.500 ε, ε, κρούσματα. πέραν τώρα της Κίνας η ε, Κόρεα, Νότιος Κορέα με περισσότερες 5.000 περιπτώσεις, η Ιταλία με 2.500 περιπτώσεις και, και το Ιράν με 2.400 περιπτώσεις είναι οι χώρες που ε, πλήττονται περισσότερο. Ε, συνολικά έχουμε 70 χώρες συνολικά από όλες τις ε, υπήρους σε διαφορετικούς βαθμούς βέβαια ε, και το κέντρο σύντηση που θα πάρει το λόγο στη συνέχεια συνεχίζει να μας ενημερώνει σε ό,τι αφορά την επιδηλωμική κατάσταση καθημερινά και δίνει και συμβουλές βέβαια στα κράτη-μέλη και στο ευρύ κοινό. Με βάση λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες του ε, ο κίνδυνος που σχετίζεται με, αυτή, με τη μόλυνση από αυτόν τον ιό θεωρείται ε, ως ε, μέτριος ο κίνδυνος έως ή και υψηλός, ανάλογα δηλαδή με τις συνέπειες ε, στην ίδια αυτού του ιού. Άρα λοιπόν, παρότι η κατάσταση δεν είναι η ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη, παρόλα αυτά ε, αυτή τη στιγμή ο ιός βρίσκεται ε, σε, στην κατάσταση του να προσπαθούμε να περιορίσουμε την διάδοσή του. Βρισκόμαστε στη φάση του κομμένου του περιορισμού, άρα δηλαδή προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους θύλακες ε, στους οποίους έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα και να ε, δούμε πώς έχει γίνει η μετάδοση. Επίσης σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε ε, ετοιμαζόμαστε ακριβώς και για το ε, χειρότερο δυνατό ε, σενάριο. Άρα λοιπόν η Επιτροπή προσπαθεί να ασκήσει πιέση στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλη ετοιμότητα και κατάλληλε υποδομέ, κατάλληλε δυνατότητε σε ό,τι αφορά την ιατρική περίθαλψη έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ένα σχετικά μεγάλο αριθμό ασθενών, για παράδειγμα υποδομέ ε, υγεία σε περίπτωση που υπάρξει ένα μεγάλο κύμα, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη αύξηση των ασθενών ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού σε αυτόν τον ε, ιό, δηλαδή οι πιο ηλικιωμένοι, αλλά και εκείνοι που πάσχουν από χρόνε ασθένειε ε, και αισθήματα υγείας. Επίσης, ε, βρισκόμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά αυτή την ετοιμότητα και αντιμετώπιση κινδύνου και να υπάρχουν και τα απαραίτητα σχέδια δράση για περίπτωση πανδημία που υποχρεούνται να έχουν τα κράτη-μέλη. Καθώς λοιπόν η Επιτροπή παρέχει όλη αυτή την υποστήριξη αλλά και οικονομική υποστήριξη και ε, υποστήριξη σε επίπεδο μελτίας, σε επίπεδο logistics, ταυτόχρονα όλες αυτές οι υπηρεσίες βέβαια υγείας παραμένουν στο, στην εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και παρότι λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή τονίζει ότι τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι ε, ανάλογα του ε, κινδύνου και να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και να αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο τη πανδημία. Θα πρέπει να είναι σε θέση να τα ε, εφαρμόσουν με ταχύ τρόπο έτσι ώστε να διακοπεί η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και έτσι να οριστή η εξάπλωση του ιού. Για παράδειγμα, μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν και αυτά είναι ενδεικτικά ε, για παράδειγμα, η αξιολόγηση των συνθήκων για την διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, ε, η πάυση λειτουργία ε, διαφορετικών εγκαταστάσεων, η διάθεση προσωπικού, εξοπλισμού προσωπικής προστασίας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, η αξιοποίηση συμπληρωματικού εργατικού δυναμικού, για παράδειγμα, συντοξιοδοτημένοι ε, ιατροί ή και φοιτητέ ιατρικής, η συγκέντρωση του απαραίτητου εξοπλισμού και του υλικού οι απαραίτητε επαφέ με του προμηθευτέ ώστε και νομικό πλαίσιο ώστε να υπάρχουν αυτέ οι προμήθειε και επίση νομικέ ε, νομικέ διατάξει ή νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να επιβληθούν μέτρα καραντίνα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι δυνατό να, να είναι στη διάθεση των κρατομελών όλα αυτά τα μέτρα, προκειμένου να ληφθούν σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί με βάση και τι ε, συμβουλέ του ECDC αλλά και ε, τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Η λήψη λοιπόν των κατάλληλων μέτρων σε αυτή τη φάση μπορεί να μας βοηθήσει να επιβραδύνουμε τη μετάδοση ή να μας δώσει περισσότερο χρόνο σε ό,τι αφορά την περαιτέρω εξέλιξη αυτών των κρουσμάτων ε, αυτού του ιού. Αυτό λοιπόν ο συμπληρωματικό χρόνο που δίνουμε στον εαυτό μα ε, είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει τη δυνατότητα σε αισθήματα υγεία να προετοιμαστούν ε, και προκειμένου να αντιμετωπίσουν ε, δηλαδή την αναμενόμενο αυξανόμενο αριθμό ασθενών και προκειμένου βέβαια να έχουν για το κατάλληλο απόθεμα σε ό,τι αφορά τα αντιϊκά φαρμακευτικά σκευάσματα. Και γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να θέσουν σε δράση από τώρα τα σχέδια ετοιμότητά του. Και επίση καλεί τα κράτη-μέλη να βρίσκονται σε επαφή με το ευρύ κοινό. Δηλαδή είναι πολύ, καλό, είναι πολύ απαραίτητο να βρίσκεται, ε, να υπάρχει ευαισθητοποίηση του ευρέω κοινού και ε, σωστή καθοδήγηση. Δηλαδή θα πρέπει να βασιζόμαστε εδώ σε δεδομένα και να μειώσουμε τι εσφαλμένε πληροφορίε και τα fake news που κυκλοφορούν. Εμεί από την πλευρά τη Επιτροπής παραμένουμε σε συνεχή επικοινωνία με τα κράτη-μέλη, χρησιμοποιώντα ε, τρία εργαλεία. Καταρχήν το σύστημα πρόορισε ε, ενημέρωσης και ετοιμότητας ε, από εκεί και μετά. Το ε, σύστημα συναντήσεων τη Επιτροπή που επιτρέπει τον συντονισμό μεταξύ όλων των ακρότων μελών και οι δυνατότητε επικοινωνία τη Επιτροπή με το ευρύ κοινό. Και, αξιοποιούμε λοιπόν αυτέ τι τρει μεθόδου ή τα τρία εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα, αν θέλετε, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τι συνέργειε που μπορούμε να έχουμε για την επαφή με το ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο λοιπόν τη ε, δυνητική εξάπλωση αυτή τη ασθένεια στο σύνολο τη Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συντονισμό των σχετικών μέτρων, συντονισμό και με τα ε, γειτονικά ε, κράτη. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να πω πω η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία μέχρι στιγμή δεν έχει προτείνει περιορισμό στο εμπόριο ή στη, σε ό,τι αφορά την το να μπορεί κανεί να ταξιδεύει. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε ε, τι ε, συμβουλέ από την πλευρά τη Παγκόσμια Παγκόσμιας Υγεία και του ECDC όπως επιβεβαιώθηκε και από του υπουργού τον Φεβρουάριο. Ε, τώρα, επιτρέψτε μου να σα ενημερώσω σε σχέση με τι τελευταίε εξελίξει. Ε, ξεκίνησε ένα διαγωνισμό από πλευρά τη Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό στο πλαίσιο δηλαδή της διαδικασία σε ό,τι αφορά τις ε, τα ιατρικά αντίμετρα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τέτοιων ε, ε, προϊόντων. Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη αυτών των προϊόντων αυτή τη στιγμή στην αγορά και έτσι θα υπάρχει δυσκολία για την κάλυψη των αναγκών όλων των κρατών μελών. Επίση, υπάρχουν μια σειρά από κοινέ δράσει που έχουμε ξεκινήσει σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την υποστήριξη των εργαστηρίων προκειμένου να προβαίνουν στι απαραίτητε δοκιμέ, αλλά και προκειμένου και στα, στη μία εισόδου στη χώρα να υπάρχουν δυνατότητε ελέγχου. Όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα και στο πρόγραμμα υγεία έχουν προβλεφθεί. Και επίση, και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά και η CDC, αλλά και ο Οργανισμό ασφάλεια ε, τη αεροπορία, έχουν προετοιμαστεί καταλήλω για την αντιμετώπιση αυτή τη κρίση. Ε, σε ό,τι αφορά την ανάγκη ε, διασφάλιση των εσωτερικών μα συνόρων, τον Φεβρουάριο οι Υπουργοί ε, της Ιταλίας αλλά και των γειτονικών χωρών συναντήθηκαν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει μια συντονισμένη απόκριση στην Ιταλία αλλά και στι γειτονικέ χώρε. Οι υπουργοί τόνισαν ότι δεν χρειάζεται να επιβληθούν έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα και δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, δηλαδή να ληφθούν μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρούνται δυσανάλογα και υπερβολικά βαριά. Οι υπουργοί θα συνεδριάσουν και πάλι αύριο, στο πλαίσιο δηλαδή σύνθεση ε, Συμβουλίου Υγείας, και εμείς ε, είμαστε κατηγορηματικά υπέρ του καλύτερου συντονισμού και των αναλογικών μέτρων. Και επίσης θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας κοινοποιήσουν τις ανάγκες τους έτσι ώστε να λάβουν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους διαφορετικούς τομείς. Ο Ιωάννης Λούκλερ, ο διευθυντής δηλαδή ε, για την διαχείριση έκτακτων ε, καταστάσεων από την Ελληνική Διεύθυνση ΕΚΟ βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μου, οπότε μπορεί να πάρει και εκείνο το λόγο αν το επιθυμείτε. Ναι, θα υπάρξουν και ερωτήσει σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα. Τώρα θα δώσω το λόγο από την Στοκόλμη στην Διευθύντρια του ECDC. Σας ευχαριστούμε πολύ που, έχετε, που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστούμε την τεχνική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και την γραμματεία που κατάφεραν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες που αφορούν και σχετίζονται με αυτήν την ε, ε, τηλεδιάσκεψη η οποία συνδέεται και με τους θαλάμους διερμηνίας αλλά και με το, το, το σύστημα web streaming. Apparently. So, uh, you very much and, uh, Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και έχετε το λόγο αγαπητή κυρία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που με προσκαλέσατε σήμερα. Θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση ε, και να σας εξηγήσω τις τελευταίες πιο πρόσφατες αξιολογήσεις ε, κινδύνου ε, που κάναμε. Ελπίζω ότι τώρα θα βλέπετε την διαφάνεια που δείχνει την επιδημονική κατάσταση στον κόσμο. Οι διερμηνείς δεν τη βλέπουν. Ε, και αυτή τη στιγμή έχουμε παραπάνω από 80.000 ε, ε, πρόεδρος. Εάν κάποιος μπορούσε να μας τα δείξει, θα ήταν πάρα πολύ καλό. please the next one. Επόμενη διαφάνεια λοιπόν. Εδώ βλέπετε την ε, κατάσταση πάνω από 95.000 ε, ε, ε, κρούσματα. Ε, εδώ με μπλε ε, βλέπετε τον πίνακα που αφορά την μετάδοση εκτός Κίνας και τις περιπτώσεις εκτός Κίνας. Βλέπουμε όλο και περισσότερες περιπτώσεις εκτός Κίνας παρά εντός. Σε τούτο το γράφημα βλέπετε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το Μόναχο, το, Σαν, το Μονακό, συγγνώμη, το, το κρατήδιο του Αγίου Μαρί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. Με κίτρινο ε, βλέπετε όλες τις ε, αναφερθήσεις ε, περιπτώσεις στην Ιταλία και διαπιστώνετε ότι την 21η Φεβρουαρίου είχε τέσσερις αναφερόμενες περιπτώσεις η Ιταλία και μέσα σε δύο εβδομάδες έχουν ξεπεράσει τώρα τις 3.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεταδοτικός είναι αυτός ο ιός. Στις προηγούμενες εβδομάδες ε, ε, αυξήθηκαν τα κρούσματα COVID-19 και στην Ιταλία και στη Γερμανία και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Και ε, τώρα οι διάφορες χώρες βρίσκονται σε διάφορες φάσεις. Έχουμε λίγες χώρες που με κανένα αναφερθέν περιστατικό και χώρες μέλη με πολλές ομάδες περιστατικών. Παρακολουθούμε λοιπόν στενά την κατάσταση καθότι ε, αυξάνονται τα κρούσματα και επομένως διαρκώς επανεξετάζουμε την κατάσταση. Έχουμε την προηγούμενη Δευτέρα ε, την πέμπτη επικαιροποιημένη ε, αξιολόγηση κινδύνου όπως ανέφερθηκε ήδη προηγουμένω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, για, το, για τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ε, ΕΑΧΑ και στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, ο κίνδυνος είναι μέσο προς ε, μεγάλο, γιατί έχουμε αυξανόμενο ρυθμό περιστατικών ε, που καταγράφονται και που δεν έχουν απαραίτητα άμεση σύνδεση με τις ε, μολυσμένες περιοχές ή με, προηγούμενες, ε, με προηγούμενα κρούσματα. Η δημιουργία κλάστερς που σχετίζονται με τον COVID-19 παρόμοια με αυτά που έχουμε στην Ιταλία αναμένονται με, κίνδυνο, με βαθμό κινδύνου μέτριο έως δυνατό και σε άλλες χώρες εκτός της Ιταλίας. Επίσης λαμβάνεται ε, υπόψη ε, αλλά ως ε, μικρός κίνδυνος η ε, διευρυμένη ας πούμε μετάδοση του ιού είτε από εσωτερικά κλάστερς είτε από εξωτερικά κρούσματα. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία μελετώνται και στα οποία έχουμε προσθέσει τα μέτρα ανταπόκρισης τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν όταν μια χώρα βρίσκεται σε σχετικό κλάστερς κλάστερ 0 ε, είναι εκεί που δεν υπάρχουν περιπτώσεις ε, και που θα πρέπει οι χώρες να δουν τα ε, σχέδια ετοιμότητας. Το κλάστερ 1 είναι το σενάριο 1 λοιπόν, όταν υπάρχει ήδη μια κατάσταση με πολλές εισαγόμενες ε, ε, περιπτώσεις και δημιουργούνται κλάστες γύρω από αυτές ε, τις περιπτώσεις. Το σενάριο 2 έχουμε σενάριο με αυξανόμενα εισαγόμενα κρούσματα και επιτόπια ευρύτερη μετάδοση στην χώρα. Σενάριο 3 είναι όπου αυτές οι εστίες, οι οποίες αρχικά ήταν ήταν αναπεριφέρεια διευρυνόμενες ε, ε, ε, εντάσσονται στην ίδια περιφέρεια και τέλος έχουμε το σενάριο το οποίο αφορά μια κατάσταση όπου έχουμε ευρεία μετάδοση και όπου τα συστήματα υγείας πλέον βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά την ετοιμότητά τους. Εκεί θα πρέπει να βρεθούν περισσότερα κρεβάτια κομμάτια μεθ ε, και να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα όσον αφορά την έλλειψη ιατρικού νοσηλευτικού ε, προσωπικού. Μπορεί να υπάρχει και έλλειψη ε, προστατευτικού ατομικού εξοπλισμού ακόμα και πρόβλημα όσον αφορά τον έλεγχο των, της ύπαρξης ιού ή όχι. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες τώρα σιγά σιγά περνάνε στο σενάριο 2. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε η Γενική Διεύθυνση Σάντε. Τώρα είναι η ώρα που θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ενεργοποιήσουν τα σχέδια ετοιμότητά τους, κυρίως όσον αφορά ε, τα, τις κλίνες τις νοσοκομιακές, καθώς επίσης ε, και το ε, νοσοκομιακό ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όσον αφορά την υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη, έχουμε κοινή ε, ομάδα από το ECDC και τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έφτασε, έφτασαν στην Ιταλία έτσι ώστε ε, να παράσχουν οποιαδήποτε δυνατή αρρωγή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επίσης, ε, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και άλλα κράτη-μέλη εάν και εφόσον μας ζητηθεί. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 60 μέλη του προσωπικού μας ε, που ασχολούνται αποκλειστικά με τον COVID-19 και έχουμε τον μέγιστο βαθμό ε, ενεργοποίησης του Κέντρου Αντιμετώπισης Κρίσεων ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου. Ε, καθημερινά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας επικαιροποίησης. Εκτός από αυτές τις ε, διαρκείς ενημερώσεις και δημοσιεύσεις, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη είτε αν προσκληθούμε και να πάμε επί είτε παρέχοντας ε, από εδώ, από μακριά, ε, μέσω βίντεο ή μέσω τηλεφώνου κάποιες ε, οδηγίες. Επίσης μπορούμε, αν μας δώσουν κάποια έγγραφα, κάποια κείμενα, να τα χτενίσουμε λίγο έτσι ώστε το μήνυμα που θα δώσουν στο κοινό να είναι πιο καθαρό. Ε, πρέπει να σας πω επίσης ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ε, στον Μητρικό Οργανισμό στην ε, ε, Γενέβη αλλά και με αντένες που έχει παντού μελετά το θέμα. Επίσης έχουμε ένα advisory forum έτσι ώστε να μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να, έχουμε, να ανταλλάσσουμε σκέψεις σχετικά με το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ε, βεβαίως εμείς διαρκώς αξιολογούμε την κατάσταση, επανεξετάζουμε, επικαιροποιούμε και τους χάρτες και όλα τα στοιχεία σε ημερήσια βάση. Επίσης στην ιστοσελίδα μας Έχουμε ένα, ε, μια έκθεση σχετικά με την απειλή ε, του COVID-19. Ε, επικαιροποιούμε τα πάντα. Αν πάτε στην ιστοσελίδα μας ε, θα έχετε πρόσβαση σε όλα από το κινητό σας τηλέφωνο. Είναι πολύ απλό. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτού δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί κλειστή συνεδρίαση με τους ε, συντονιστές ε, και την ε, Επίτροπο, την κυρία Κυριακίδη, που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Θα έχουμε συζήτηση όμως με τους συντονιστές και εκείνη την Πέμπτη πάνω στον κοροναϊό. Ο κύριος Σελίζε, Τούτελαντ. Παύλης, Madame Rondinelli. Wow, wow, wow. Okay, so one, two, three, four, five, six more. Okay. So we close the list. Perfect. Let's... Κλείνουμε το κατάλογο των ομιλητών και ξεκινάμε από τον Πέτερ Λίζα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευχαριστώ και την κυρία Άμονα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Γιατρός είμαι και όταν μιλώ με συναδέρφους ειδικού στους ιούς, δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς απαντήσεις, γι' αυτό δεν ζηλεύω κανένα που πρέπει να πάρει αποφάσεις αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ε, παραμείνουμε ήρεμοι, να μην πανικοβληθούμε. Αλλά βέβαια το να πει κανεί μην πανικοβληθεί είναι ο καλύτερο τρόπο να προκαλέσει κανεί πανικό. Να παραμείνουμε λοιπόν ψύχρεμοι. Υπάρχουν αρρώστιες που σκοτώνουν πολλούς ε, ανθρώπους ε, κάθε μέρα, ε, άλλες ασθένειες, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να επαγρυπνούμε και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω την πρώτη επίκριση στου δύο μιλητές μας. Τα δεδομένα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαφέρουν ε, από αυτά που μας έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Πρόληψης και αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται. Ο ένας είπε 3.400 θανάτους, άλλος είπε 4.200. Δεν επιτρέπεται να μην συμφωνούν τα στοιχεία μεταξύ τους. Και θα πω κάτι που θα σας ανησυχήσει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ε, γνωρίζουμε την κατάσταση. Κανένα από τα δύο νούμερα αυτά δεν ισχύει. Ε, έχουμε πολύ περισσότερες περιπτώσεις στην Ευρώπη, απλά δεν έχει γίνει η διάγνωση. Και δυστυχώς στην Ιταλία είχαμε 100 θανάτους. Και αν θεωρήσουμε ότι, ε, ότι δόξα το Θεό αυτός ο ιός δεν είναι τόσο ε, ε, θανατηφόρος και ότι το 0,2% όσων ε, ε, ε, προσβάλλονται από τον ιό πεθαίνουν, τότε σημαίνει ότι θα έχουμε τουλάχιστον χίλιες περιπτώσεις στην Ιταλία και στη δική μου χώρα, την Γερμανία, Έχουμε παραπάνω από τις 200 περιπτώσεις που έχουν ε, αναφερθεί. Δεν ε, πιστεύω ότι ο καθένας που ε, φταρνίζεται θα πρέπει να εξετάζεται, αλλά τουλάχιστον όποιος έχει πυρετό θα πρέπει να εξετάζεται. Προβλήματα στα πνευμόνια δημιουργεί ο κοροναϊός, όχι απλό κρυολόγημα. Θα πρέπει λοιπόν έτσι να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και την ε, εξάπλωση της ασθένειας δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε, μπορούμε όμως να την ε, περιορίσουμε σημαντικά. Βλέπουμε προσπάθειες ε, να περιοριστεί η δημόσια ζωή στην Ευρώπη. Είδαμε τα μέτρα του Προέδρου Σασόλη. Δεν έφερα καμιά αντίρρηση να περιορίσουμε κάπως ε, τις ε, μη ε, απαραίτητες μετακινήσεις, το βρίσκω λογικό. Και με όλη την εκτίμηση και με όλο το σεβασμό βρήκα κάπως οριακή την εκθεσινή εκδήλωση με την Γκρέτα θα γίνει η Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Συζητιέται αυτό. Δεν ε, θα ήθελα εγώ να λάβω απόφαση. Αν όμως πραγματοποιηθεί η Ολομέλεια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν ε, γίνει διάγνωση κάποιου όταν θα βρίσκεται στη, στο Στρασβούργο, θα πρέπει να ε, εφαρμόσουμε κάποιο σχέδιο ώστε να μην χωρίσουμε τους ανθρώπους από τις οικογένειές τους, να μπορούν δηλαδή να πάνε για καραντίνα στο σπίτι τους και όχι στο Στρασβούργο. Και αυτό είναι ισχύει για όλους. Ε, για φανταστείτε τώρα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να κολλήσει στην Ιταλία και να μπει σε καραντίνα. Θα πρέπει τουλάχιστον να μπορεί να μπει σε καραντίνα στι Βρυξέλλες και να συνεχίσει τη δουλειά τη. Πολύ σύντομα όσον αφορά τα πολιτι... τις πολιτικές εκκλήσεις. Περιορισμένο χρόνο έχω, ο Πρόεδρος ε, σίγουρα έχει δίκιο. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη όσον αφορά τον συντονισμό. Οι συστάσεις ε, δεν διαφέρουν. Ε, γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιορισμένες νομικές δυνατότητες, αλλά πολιτικά θα πρέπει να ε, λάβουμε πολύ πιο στεναρή θέση, να υποβάλουμε συστάσεις, να συνεργαστούμε πολύ στενά μεταξύ μας, για παράδειγμα όσον αφορά τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις ε, θεραπείες. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πετύχουμε από κοινού ε, μαζί καλά αποτελέσματα. Θα μπορούσα να μακρηγορήσω, αλλά κοιτάω και το ρολόι. Πρόεδρος, ε, σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς για το που θα πραγματοποιηθεί η Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Πρώτον. Και δεύτερον, σας παρακαλώ να περιοριστείτε στον χρόνο ομιλίας σας για να ε, προλάβουν όλοι να πάρουν το λόγο. Η Γιούτε Κούτελαντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και την δόκτωρα Άμον ε, από το ECDC για την ε, πολύ καλή εισήγησή της. Είναι σημαντικό να παραμένουμε ενήμεροι και να κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να φροντίσουμε όλοι να είναι σωστά ενημερωμένοι και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι Υπουργοί Υγείας να μπορούν να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποτρέψουμε ε, τη μετάδοση της νόσου και σε περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα να έχουμε και αποτελεσματικά συστήματα υγείας ε, που να κάνουν σωστή αξιολόγηση και να λαμβάνουν σωστά μέτρα. Επίσης, η εφαρμογή της καραντίνας θα πρέπει να γίνεται με καλό τρόπο ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι αναλογικό μέτρο να ε, παραμείνουν οι άνθρωποι σπίτι τους σε περίπτωση που έχουν ε, ε, κολλήσει τον ιό. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Πέτερ ότι είναι σημαντικό να μην τα στοιχεία, ε, να μην υπάρχουν ε, διαφορές ε, όσον αφορά τα στοιχεία που δημοσιεύονται. Επίσης, όσον αφορά τον χρόνο επόασης, αρχικά είχε υποθεί ότι είναι δύο εβδομάδες, ενώ αργότερα υπήρξαν αμφιβολίες σχετικά με αυτό. Νομίζω ότι ακόμα και όταν υπάρχουν αμφιβολίες, ε, ακόμα και αυτές ε, είναι καλό να ε, είναι σαφείς. Ακόμα και εμπειρογνώμονες είχαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήταν ασαφής. Νομίζω ότι καλύτερα να πει κανείς εάν δεν είναι βέβαιος παρά να, είναι, να φανεί απολύτως βέβαιος και κατόπιν να αλλάξουν τα στοιχεία. Εγώ θέλω οι άνθρωποι στην Ευρώπη να νιώθουν ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε την εξάπλωση του ιού και όχι απλά να αντιδρούμε όταν κάποιος ήδη έχει πληγεί από τον κοροναϊό. βλέπουμε για παράδειγμα να κλείνουν σχολεία σε περιπτώσεις που ίσως ε, να μην είναι απαραίτητο. Θα ήθελαμε λοιπόν ε, συμβουλές σχετικά με τα προληπτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να περιορίσουμε την ε, εξάπλωση του ιού, διότι... Και ναι, ναι, κλείνω μπορεί να ε, ε, αυξάνεται ο κίνδυνος ε, εάν δεν κλείνουν επιχειρήσεις και ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να περιορίσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στεφανούτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ για αυτές τις παρουσιάσεις. Γνωρίζουμε πως το ECDC επιλαμβάνεται διαφορετικών ζητημάτων, αλλά ίσως ε, να μην είναι αρμοδιότητα του το ερώτημα που θα θέσω, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να το θέσω. Ποια είναι στα στατιστικά σχέδια της Επιτροπής σε ό,τι αφορά ε, τις ε, προμήθειες σε φαρμακευτικά σκευάσματα και σε εξοπλισμό ε, προσωπικής προστασίας γιατί σίγουρα η κατάσταση ε, είναι πολύ διαφορετική ανά κράτος μέλος και δεν θα πρέπει να χρειάζεται κανείς να ζητιανέψει το εισαγωγικών από την γειτονική του χώρα ε, τέτοιου είδου εξοπλισμό. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα, καθώς ίσως να χρειαστεί βέβαια και κάποια στιγμή τα σύνορα να κλείσουν. Οπότε υπάρχει τέτοιο σχέδιο και ποιο είναι αυτό, πώς είναι διαμορφωμένο. Επίσης ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ε, ακριβώς είναι αυτό το app στο οποίο αναφερθήκατε. Ε, αυτά τα δεδομένα που περιλαμβάνει ισχύουν για όλα, είναι διαθέσιμα και όλα τα κράτη-μέλη. IND. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έγινε λόγο για την, έγινε για την Ιταλία και για το βαθμό επιμόλυνσης που έχουμε. Η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών που με διαφάνεια δόθηκαν πραγματικά στοιχεία ε, σχετικά με τα περιστατικά τα ε, σημερινά. Ε, ενδεχομένως και λέω ενδεχομένως αυτό δεν έγινε στα άλλα κράτη. Αυτό έχει επίπτωση όχι μονάχα σε επίπεδο, διαφάνει, ε, σε επίπεδο διαχείρισης της ψύχωσης που σχετίζεται με τον ιό αλλά και έχει οικονομικές επιπτώσεις Κοιτάξτε, εδώ και μέρες έχουν ε, υπάρξει πολλά ε, αιτήματα ε, που ζητούν από διάφορες αλυσίδες διανομής που ζητούν παράλογες διασφαλίσεις από την Ιταλία. Επίσης υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ζητάνε να υπάρχει μια ετικέτα corona free, coronavirus free σε όλα τα προϊόντα. Αυτά όμως είναι πολύ κακά πράγματα και εν πάση περιπτώσει ε, δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Made in Italy που είναι ένα μπραντ πολύ σημαντικό για την Ιταλία και σκυλεύονται στην ουσία την Ιταλική οικονομία ε, ε, λόγω μιας κατάστασης που επικρατεί τώρα. Εγώ θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτες τέτοιες αιτήσει επιπλέον πιστοποίησης και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τεθούμε απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και που στην ουσία είναι ε, προσπάθεια εγχειρηματοποίησης της κατάστασης και μπλοκαρίσματος των Ιταλικών εξαγωγών. Ε, δεν υπάρχει επίσης ε, καμία επιστημονική τεκμηρίωση που να λέει ότι μέσω των τροφίμων μπορεί να μεταδοθεί το ο ιός. Ευχαριστώ. κυρία Παύλος από τους Πρασίνους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και σας ευχαριστούμε που μας λέτε ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν από τα κράτη-μέλη ε, ασχέτως εάν ε, ε, τους έχει ζητηθεί ή όχι. Συμφωνώ ε, με αυτήν την αξιολόγηση για την περίπτωση της Ιταλίας, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες ε, επιπλέον περιπτώσεις τις οποίες και κρούσματα που όμως δεν έχουν καταγραφεί γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται τα καλά, είτε γιατί δεν θέλουν ε, να πάνε στον ε, γιατρό ή δεν έχουν καθόλου ε, συμπτώματα ή συμπτώματα τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως σχετιζόμενα με τον ιό. Είναι, είναι βέβαιο ότι πρέπει να έχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη πολύ περισσότερα από τα δηλωμένα. Ε, ας πούμε από την άλλη μεριά μπορεί να ελέγξουμε ανθρώπους που έχουν πνευμονικά προβλήματα αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι ε, ε, έχουν έρθει σε επαφή με άλλους οι επιδημιολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι λένε ότι τα, ε, ε, το υλικό ε, φορτίο το οποίο μπορεί να είναι στον Φάριγκα μπορεί να μην κατέβει ή να μην έχει κατέβει ακόμα στους πνεύμονες. Δηλαδή μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν συμπτώματα αλλά ασυμπτωματικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν ήδη υλικό Um, Έχουν ήδη οικό στους ε, φάριγγες, ε, στον φάριγγα. Εν πάση περιπτώσει όμως η πραγματική μου ερώτηση είναι η εξής. Ε. υπάρχουν συγκεκριμένες ε, συμβουλές ε, για αυτούς που ας πούμε ζουν μόνοι τους ε, ή που δεν έχουν κάποιον να τους προσέχει, τι γίνεται με τους ασυμπτωματικούς, τι γίνεται με τους άστεγους που ζουν στο δρόμο και που έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αρπάξουν τον ιό γιατί έρχονται πολύ σε επαφή με κόσμο, δεν πλένονται ικανοποιητικά, δεν απολυμένονται καθόλου. Επίσης, ε, σε μέρη όπως η Λέσβος, ας πούμε, όπου έχουμε ε, ε, κέντρα υποδοχής για τρεις, που έχουν χτιστεί για 3.000 ανθρώπους και αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολλές χιλιάδες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Τι γίνεται εκεί. γιατί ε, όντως θα μπορούσε να υπάρξει πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη μετάδοση. Από το ECR, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει το άρθρο 168 της Συνθήκης Λειτουργίας που ε, αναφέρει σαφώς ότι τα κράτη-μέλη είναι ε, υπεύθυνα και έχουν ε, απόλυτη ευθύνη και αρμοδιότητα για τις υπηρεσίες υγείας και την οργάνωσή τους. Όσον αφορά δε, τα προγράμματα και σχέδια ετοιμότητας, ναι, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να αυξήσουν την ικανότητα υποδοχής ασθενών και την, τα προγράμματα πρόληψης ε, ε, λοιμόξεων. Πρέπει λοιπόν να ετοιμαστούμε για τα ε, επόμενα βήματα και για τα επόμενα σενάρια έτσι όπως τα δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το ECDC κυρίως για το σενάριο υπαριθμών 4. Είναι τέτοιο το σενάριο όπου ενδεχομένως να ξεπεραστεί το σύστημα υγείας από τις αιτήσει συνδρομής και από τους ασθενείς. Επίσης ε, δεν υπάρχει διαγνωστικό τεστ ε, στην ε, διαθέσιμο στην αγορά. Το πρόβλημα θα μπορούσε να αυξηθεί υπερβολικά. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Σύμφωνα με την Κομισιόν ε, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει ε, τέτοιο πρόβλημα τόσο μεγάλο ώστε να έχουμε πραγματική έλλειψη φαρμάκων ε, και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βοηθήσει την αλυσίδα προμήθειας των φαρμάκων εάν προχωρήσει τόσο πολύ και εξαπλωθεί ο ιός. Επίσης, ποια είναι τα σχέδια ε, καταπολέμησης ε, ε, των περιπτώσεων κατάχρηση ανταγωνισμού όπου ο καθένας παίρνει ό,τι φάρμακο βρει και δεν τηρούνται οι κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά γίνονται για να προλάβουμε την εξάπλωση του κοροναϊού, αλλά ε, εγώ νομίζω ότι δεν γίνονται αρκετά για να αποτρέψουμε ε, μελλοντικές εμφανίσεις νόσων όπως είναι ο εμπόλα, γρήπη, SARS ε, και άλλες ε, ασθένειες που προκαλούνται από νυχτερίδες, πουλιά, πρόβατα κλπ. ε, αυτός ο κοροναϊός ε, εξαπλώθηκε ε, από ζώο σε ζώο μέχρι να ε, φτάσει τον άνθρωπο. Και ο τρόπος που χειριζόμαστε τα ζώα έχει σημαντικές συνέπειες. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερώτηση τι θα κάνει στο μέλλον για να προλάβει τέτοιες περιπτώσεις. Ε, θα εφαρμόσουμε καλύτερους κανόνες όσον αφορά τα ζώα από ότι οι Κινέζοι. Επίσης, ε, έχουν ακουστεί κάποια κρούσματα στο Μεξικό. Μήπως θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό τώρα και όχι να περιμένουμε. Επίσης, όσον αφορά το εμπόριο ε, των ζώων ε, υπάρχουν εδώ και κάποιες ε, αρνητικές ε, συνέπειες από την απαγόρευση. Είδαμε τόσα κουφάρια ζώων από την Βουχάν. Έχετε ακούσει κάτι σχετικό. Ευχαριστώ. Από το Έλκι κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη σημαντική αυτή εισήγηση. Δύο ερωτήσεις έχω με ενδιέφεραν ε, τα, πολύ τα τέσσερα σενάρια που ακούσαμε από το Κέντρο Προλήψεως Νόσων. Ε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε το σενάριο 4 ή είναι αναπόφευκτο και απλά πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε τώρα. Αυτό δεν κατάλαβα καλά. Και δεύτερον, Ακούστηκαν διάφορες υποθέσεις ε, σχετικά με την ε, πηγή ε, των, της νόσου αυτής. Κάποιοι επέστρεψαν από την Ιταλία στην Ιρλανδία, κάποιος είχε βάρδια σε σταθμό πρώτων βοηθειών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, είναι πρόβλημα και φυσικά κανένας δεν θέλει να, πανικοβα... να πανικοβληθούμε. Ε, στην ε, Καλιφόρνια όμως μόλις προκυρήθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να λάβουν αποφάσεις και γι' αυτό ακριβώς εκτιμώ αυτή την σημερινή συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες και θα αφήσουμε να μας καθοδηγήσετε. Ευχαριστώ το S&D. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ιατρός είμαι. Ε, στα επίγοντα περιστατικά και ε, θεωρώ ε, πως είναι μόνο ζήτημα χρόνου μέχρι να θεωρηθεί πλέον αυτή η κατάσταση ως ε, πανδημία, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα εδώ. Ε, ο αριθμό δηλαδή των κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεκαπλασιαστεί και ακούσαμε από το CDC τα διαφορετικά σενάρια, οπότε θα ήθελα και εγώ ε, να ρωτήσω ε, τι ακριβώς θα γίνει, γιατί προφανώς πρέπει να προστατεύσουμε τη ζωή όλων και κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Ποια είναι λοιπόν τα προληπτικά μέτρα ακριβώς που πρέπει να ληφθούν. Από εκεί και μετά αναφέρεται ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εκδηλώσεις, δημόσιες εκδηλώσεις ε, ε, ε, γιατί με αυτόν τον τρόπο υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης αλλά για παράδειγμα όλες οι αστικές μεταφορές μικρών αποστάσεων τα σχολεία και ό,τι καθεξής συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά δεν υπάρχει κανένας είδους καραντίνα όπως για παράδειγμα έχει εφαρμοστεί στην Ιαπωνία εάν πραγματικά βρεθούμε σε κατάσταση ε, πανδημίας ε, θα προκύψει το ζήτημα όχι μόνο ε, εκείνο που ασθενούν αλλά και το γεγονός ότι ακριβώς υπάρχει, θα υπάρχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα πλέον του ιού και τα νοσοκομεία μας και γενικά οι καταστάσεις υγείας δεν είναι αρκούντως προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Και μας είπατε ότι ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις όπου οι, ακριβώς αυτές οι, οι, οι δυνατότητες σε επίπεδο ιατρική περίθαλψη των κρατό μελών δεν θα ε, είναι επαρκή. Οπότε θα πρέπει ενδεχομένω εδώ να υπάρξει υποστήριξη και ενεργοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε για παράδειγμα να γίνουν από τώρα εισαγωγέ σε ό,τι αφορά φαρμακευτικά συσκευάσματα και προστατευτικό εξοπλισμό. Και ε, στην περίπτωση, για παράδειγμα, που πραγματικά βρεθούμε στο σενάριο 4, πώ θα έχουν εκεί τα πράγματα, θα υπάρχει πραγματικά κάποια δυνατότητα να έχουμε προμήθεια αυτών των φαρμάκων και αυτού του εξοπλισμού. Ευχαριστώ ο κύριος Βοτζακ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα συμφωνήσω με αυτά που υπόθηκαν ήδη, δηλαδή ας είμαστε προσεκτικοί, ας μην εσείς πανικός και εγώ θα ήθελα να θέσω στην ατρό δύο ερωτήματα. Καταρχήν, το ζήτημα της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των δεδομένων που προερχόνται από την Κίνα. Αυτό το είχαμε συζητήσει την τελευταία φορά εδώ καθώς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά το κατά πόσο εμπιστευόμαστε τα δεδομένα που έρχονται από την Κίνα. Δηλαδή μπορούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που μας διαβιβάζει αυτή η χώρα από τη μία μέρα στην άλλη. Και βέβαια τίθεται και ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και των δικών μας δεδομένων. Από εκεί και μετά ένα δεύτερο ερώτημα είναι ε, το κατά πόσο πραγματικά υπάρχει ανάπτυξη ενό αποτελεσματικού φαρμάκου, γιατί ακούσαμε κάτι ότι υπάρχει ε, κάτι τέτοιο στις, στις, ε, στο Πολιτείες. από εκεί και μετά, ένα τρίτο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω είναι ο προστατευτικό εξοπλισμό για τον οποίο ήδη υπάρχει έλλειψη σε ό,τι αφορά το ίδιο το ιατρικό προσωπικό. Θα πρέπει δηλαδή να απαγορεύσουμε την εξαγωγή τέτοιου εξοπλισμού προ το παρόν. Στη δική μα ε, χώρα το έχουμε ήδη κάνει, οπότε νομίζω πω θα πρέπει να σκεφτούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμπληρωματικά μέτρα. Γιατί σε διαφορετική ε, περίπτωση δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο για την ανάπτυξη και ενό εμβολίου, όπω ε, είπε και ο κύριο Πετρελίζη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ όλους όσοι εργάζονται ε, πάνω στο θέμα αυτό ε, και βεβαίως μεγάλος ο προβληματισμός, είναι λογικό αυτό και εν μέρη και ο πανικός που προκαλείται ε, στον κόσμο, στους πολίτες μας από αυτόν τον ιό είναι ανθρώπινο. Ωστόσο η πολιτική θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της βασιζόμενη στην επιστήμη και στα επιστημονικά στοιχεία, έτσι όπως υπόθηκε και προηγουμένω από τους έγκριτους εισηγητές μας. Η πρόεδρο Βοντερ Λάγεν είπε ότι θα θεσμοθετηθεί μία task force ε, και ότι ήδη από τις 13 Φεβρουαρίου δουλεύει η Ευρώπη πάνω στο θέμα αυτό. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι άργησε. Άργησε διότι τα νέα τα οποία είχαμε για τον ιό αυτό ε, ήδη κυκλοφορούσαν από μήνες και για μία ακόμα φορά εγώ που είμαι πεπισμένη φιλοευρωπαία ε, και που είμαι πάντα φανατικά υπέρ της Ευρώπης ε, λέω ότι αργήσαμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δουλέψουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερο το λέω γιατί οι πόροι αν ε, δεν κάνω λάθος, 230 εκατομμύρια αναρωτιέμαι και σας ρωτώ και εσείς, ε, είναι άραγε ε, αρκετά, πρέπει να αυξηθεί αυτή η χρηματοδότηση, η έρευνα επίσης για το εμβόλιο, ήδη έχουν δοθεί 20 εκατομμύρια, είναι αρκετά, πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους για την έρευνα που είναι θεμελιώδους σημασίας και για την προκείμενη περίπτωση. Δεν μπαίνουμε τώρα στην ουσία των πόρων που θα πρέπει να δώσει η Ευρώπη όσον αφορά την οικονομία, γιατί χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, ε, είναι χώρες ε, οι οποίες αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την κινητήρια δύναμη της Ευρώπης και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα και όσον αφορά αυτό το θέμα. Για την Ιταλία, εγώ είμαι Ιταλία και είμαι περήφανη ε, για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μου και ο υπουργό υγεία διαχειρίστηκαν το θέμα. Όμως, όμως η Ιταλία ίσως να έκανε αυτό που δεν έκαναν άλλε χώρε, Εγώ συμφωνώ με τον Πίτερ Λίζε. Είναι πολύ περισσότερες ε, οι ε, περιπτώσει στην Ευρώπη. Δεν τις γνωρίζουμε. Εμείς λέμε ότι είναι τόσα πολλά τα κρούσματα γιατί κάναμε buffer zones, γιατί αποκλείσαμε περιοχές ολόκληρες. Επομένως, το θέμα αυτό της γρήγορης και προφανούς ε, μετάδοσης του ιού δεν μπορεί να αφορά μονάχα μία χώρα, θα αφορά και τις άλλες χώρες. Και αν παίρνουμε μέτρα θα πρέπει είτε όλοι να τα πάρουμε με τον ίδιο τρόπο και άλλωστε η Ευρώπη ε, αυτά τα κοινά μέτρα θα πρέπει να σκηνοθετήσει ή διαφορετικά ε, δεν έχει και πολλή έννοια γιατί οι άνθρωποι κυκλοφορούν, μετακινούνται και επομένως μεταδίδεται και ο ιός. Επομένως, πιστεύω πιστεύω ότι η Κομισιόν ε, ε, ε, και η δικιά μας και η Επιτροπή Πρόεδρε θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσει κάποιες ενδείξεις και για την επόμενη Ολομέλεια, γιατί το να μεταφέρουμε πάνω από 5.000 ανθρώπους την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ίσως είναι ένα κίνδυνο τον οποίο δεν πρέπει να επιτρέψουμε ε, να ε, ε, υπάρξει. Uh, Πρόεδρο, ε, ας αφήσουμε τα αρμόδια όργανα να πάρουν τις αποφάσεις τους. Παρακαλώ πολύ, επόμενος ομιλητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ως Ιταλίδα δεν μπορώ παρά να εκφράσω τον προβληματισμό όλων μας και ολόκληρης της Ευρώπης για αυτό ε, τον ε, ιό που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ε, μεταδοτικότητα καθώς επίσης και μεγάλο ρυθμό ασυμπτωματικών ασθενών. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερος. Στην πραγματικότητα ε, ε, διαπιστώνουμε πραγματική έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών κατά την άποψή μου όσον αφορά αυτή την επίγουσα κατάσταση. Όλοι γνωρίζουμε ότι το, η υγεία είναι ένα συγκεκριμένο θέμα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και όπου η επικουρικότητα έχει συγκεκριμένο εύρος. Από την άλλη μεριά είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, λείπουν τα ελάχιστα ε, ε, μέτρα τα οποία θα είναι υποχρεωτικά για όλους έτσι ώστε να συγκρατήσουμε την επιδημία και δεν θέλουμε, θέλουμε να συγκρατήσουμε την επιδημία έτσι ώστε να μην γίνει πανδημία. Ε, θα, ε, έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά είναι κυρίως όχι ερωτήσεις, αλλά ε, αιτήματα. Πρώτον, ανταλλαγή ε, πληροφοριών για τις ε, βέλτιστες πρακτικές. Δεν είναι αρκετή η ανταλλαγή πληροφοριών. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, στην χώρα μου έχουν γίνει 30.000 buffer zones ζώνες ε, αποκλεισμού και έχουμε σχεδόν 3.800 ασθενείς ε, που είτε έχουν νοσήσει είτε όχι, δηλαδή είτε είναι ασυμπτωματικοί είτε όχι. Υπάρχουν όμως άλλες χώρες ε, όπου το, ε, τα, επίσημα στοιχεία αφορούν μονάχα τους ανθρώπους, του ασθενείς που έχουν παρουσιάσει πλέον τα συμπτώματα που έχουν νοσήσει. Άρα ακόμα και όσον αφορά τι πληροφορίε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δίνουμε όλοι και ανταλλάσσουμε τις παρόμοιε και σωστέ πληροφορίε. Κι άλλο ένα αίτημα. Πρέπει να ξεκινήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα κοινό πρωτόκολλο ε, καταγραφής ε, των κρουσμάτων. Πραγματικά δηλαδή αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά τα κρούσματα και να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε ε, και την επίγουσα κατάσταση όσον αφορά την, ε, την επιμόλυνση και όσον αφορά την ε, η αντιμετώπιση υγείας. Γιατί ναι, είναι κρίσιμη κατάσταση, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε Λυπούμε που το λέω, αλλά ε, ο ιός αυτός θα οδηγήσει οπωσδήποτε και πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και την Ευρώπη εν τέλει στο σύνολό της, ε, σε μια οικονομική υποχώρηση. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν και κάποια προσήκοντα ή οικονομικά μέτρα. Ευχαριστώ. Thank you very much. So... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στη Στοκχόλμη, στο ECDC και ρωτώ ε, τι γίνεται με τη διερμηνία, αν μπορούμε να συνεχίσουμε για 5-7 λεπτά ακόμη, διότι μας τελειώνει ο χρόνος. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στο ECDC. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που μας θέσατε πολλές από τις ερωτήσεις που σχετίζονται με ε, τα δεδομένα και ε, με τους αριθμούς και τις ε, διαφορές στα στοιχεία. Εμείς λαμβάνουμε συνέχεια αναφορές. Η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία. Δεν θα εκπλήξει κανέναν ότι υπάρχουν κάποιες ελαφρές διαφορές. Αυτές οι ελαφρές διαφορές όμως δεν θα πρέπει να είναι η βασική ανησυχία. Υπόθηκε ότι ο, αριθμ, ο πραγματικός αριθμός ε, είναι μεγαλύτερος ε, από αυτούς που αναφέρθηκε. Αυτό ισχύει για κάθε ασθένεια, ιδιαίτερα για αυτές όπου η πλειοψηφία των ε, αρρώστων έχουν πολύ ελαφρά συμπτώματα και μπορεί να μην πάνε στο γιατρό. Έχουμε κοινό πρωτόκολλο παρακολούθησης ε, από τα τέλη Ιανουαρίου. Το πρωτόκολλο για την υποβολή αναφορών ε, ισχύει εδώ και κάποιες εβδομάδες και το προσαρμόζουμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους στα κράτη-μέλη σε συνεχή βάση. Αναφέρθηκε ότι όσοι δεν έχουν συμπτώματα μπορούν να μεταδώσουν την νόσο. Δεν έχουμε ε, σχετικά στοιχεία, αλλά γνωρίζουμε ότι ακόμη και τα ελαφρά συμπτώματα μπορούν να οδηγήσουν σε μετάδοση της νόσου. Οι υποθέσεις ε, αρχικά όπου ε, θεωρήθηκε ότι κάποιος δεν έχει συμπτώματα αποδείχθηκε ότι ήταν περιπτώσεις με πολύ ελαφρά συμπτώματα. Όσον αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης, ε, συνομιλούμε με τις αρχές στα κράτη-μέλη. για να διευρύνουμε τις δοκιμές και να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα του κάθε κράτους μέλους ε, για την παρακολούθηση της γρήπης ε, και για τον νέο αυτόν ιό. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Τέθηκε ερώτηση σχετικά με τα σενάρια και αν μπορούμε να αποφύγουμε να περάσουμε στο σενάριο 4. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε αυτό τελείως, αλλά όλες οι προσπάθειες που γίνονται τώρα και από τις υπηρεσίες υγείας σε τοπικό, ε, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στα κράτη-μέλη προσπαθούν να εντοπίζουν εγκαίρως τα περιστατικά, να έρχονται σε επαφή με ε, ανθρώπους ε, που θα ενεργήσουν ως ε, σύνδεσμοι και να ε, επιβραδύνουν την εξάπλωση ώστε να μην έχουμε μια άμεση όξυνση αλλά να έχουμε μια πιο ευρία καμπύλη, κάτι που θα ανακουφίσει και τα συστήματα υγείας. Με ρωτήσατε σχετικά με την ε, εφαρμογή του τηλεφώνου. Λέγεται ECDC Threat Report. Και η καθημερινή ε, ενημέρωση ε, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή αυτή. Μπορείτε λοιπόν πάντα να βρίσκετε τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Όσον αφορά ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, είναι κάτι που συζητάμε όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι σε ένα μέρος, υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδοθεί πολύ εύκολα ο ιός. Εξελίσσεται η κατάσταση και με τους πρόσφυγες, οπότε φυσικά θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτή την πτυχή. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, όσον αφορά τις ε, προβολές ε, από τους θανάτους που είχαμε μέχρι τώρα ε, όσον αφορά τον αριθμό των ε, ε, αριθμό περιστατικών, διότι το ποσοστό θνησιμότητας ποικίλει ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα και ανάλογα με την φάση της ασθένειας. Αυτό το διαπιστώσαμε και στην Κίνα. Ε, στην ε, πρώτη φάση της ε, εμφάνισης της νόσου, στη μεσαία φάση και στην τελική φάση διαφέρει πολύ το ποσοστό θνησιμότητας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά προβλέψεις. Αλλά φυσικά είναι σαφές ότι έχουμε περισσότερες υποθέσεις, περισσότερα κρούσματα από αυτά που αναφέρονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά Γενική Διεύθυνση Υγείας. Λίγες παρατηρήσεις επειδή έχει προχωρήσει ο χρόνος. Όπω σα είπα, νομίζω ότι το Συμβουλίο Υπουργών θα ασχοληθεί περισσότερο με τις επόμενες ε, φάσεις. Ε, ε, το θέμα είναι να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας ώστε να είναι προετοιμασμένα για ό,τι συμβεί στο μέλλον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εντοπίσει τις ανάγκες στα κράτη-μέλη και όσον αφορά τον εξοπλισμό και όσον αφορά τρόπους κινητοποίησης του συστήματος υγείας, όσον αφορά το θέμα της επιστοποίησης προϊόντων από την Ιταλία. Ε, εμείς δεν έχουμε ακούσει να λαμβάνονται μέτρα από άλλα κράτη-μέλη όσον αφορά την εξαγωγή αγαθών από την Ιταλία. Όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες και τους ε, μετανάστες, ε, σκοπεύουμε σε συνεργασία με τις κοινότητες και τα κράτη-μέλη να ε, εστιάσουμε ιδιαίτερα στις ευάλωτε ομάδες και φυσικά έχουμε μια ειδική κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση και στα κράτη-μέλη και στα ε, κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τα hot spots. Σκοπός είναι να μπορέσουμε να εντοπίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τα κρούσματα και να τα αντιμετωπίσουμε. Επίσης, ε, τέτοια ερώτηση σχετικά με την ε, πολιτική όσον αφορά τα φάρμακα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την αλυσίδα τροφοδοσίας, ε, διότι πολλά προϊόντα προέρχονται από την Κίνα. Επίσης και από την Ινδία, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την φαρμακευτική βιομηχανία και με τον Οργανισμό Φαρμάκων και παρακολουθούμε τις εξελίξεις για να δούμε αν υπάρξει κάτι που να απειλεί την ασφάλεια τροφοδοσίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ε, ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων και, ε, την έρευνα, 100 εκατομμύρια ευρώ έχει επενδύσει τις τελευταίες εβδομάδες ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων. κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τον ε, προσωπικό εξοπλισμό. Ε, ε, έχουμε πρόσκληση υποβολής προσφορών σε 20 κράτη-μέλη για την προμήθεια τέτοιων προϊόντων και τα κράτη-μέλη και σε εθνικό επίπεδο συναπτούν δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ε, έχει ε, αποθαρρύνει ε, τις χώρες από την εφαρμογή απαγόρευσης εισόδου-εξόδου από τη χώρα, διότι έχουν αποδειχθεί μη αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ, κυρία Διευθυντά, από την Στοχόλμη. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ε, και άλλες ευκαιρίες να, να συζητήσουμε τον κοροναϊό. Και όπως σας είπα θα έχουμε και κλεισμένο το θυρών ε, συζήτηση με τον Επίτροπο και τους ε, συντονιστές την επόμενη εβδομάδα, 18 και 19 Μαρτίου.